Καλημέρα σας. Έχουμε πάρα πολλά θέματα να συζητήσουμε σήμερα. Έτσι λοιπόν, να, να σας πω ότι έχουμε και μετάδοση από την τηλεόραση, την ιστορική τηλεόραση. Λοιπόν, για τις αποφάσεις που θετήθηκαν ε, χθες το απόγευμα από τους συντονιστές, ε, θα σας ενημερώσω. Καταρχήν, αποφασίστηκε να μην δοθεί συνέχεια στην πρόταση της τροποποίησης του κανονισμού που παρουσιάστηκε τον κύριο Σπερονή σύμφωνα με το άρθρο 2.12 που ήθελε να βάλουμε το άρθρο 49α στον κανονισμό σε ό,τι αφορά τις ε, διοργανικές συμφωνίες με το Συμβούλιο. Επιβεβαιώθηκε ο διορισμός του κ. Εφνέρ για τις, 15 ε, ε, Μαρτίου 2012 για την ε, διοργανική συμφωνία σε σχέση με τη ε, διαβίβαση εμπιστευτικών πληροφοριών στο Κοινοβούλιο από το Συμβούλιο για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας. σε ό,τι αφορά την έκθεση Φερσκόφσκι για το άρθρο 123 σε σχέση με τις γραπτές δηλώσεις διευρύνθηκε το ζήτημα βάσει τροπολογίας του κυρίου Γκολτιέρη που αναφέρθηκε και από τον εισηγητή, έτσι ώστε να συμπεριληφθεί και το θέμα των νομοθετικών πρωτοβουλειών. Επαφασίστηκε, προτείνεται να μην εκπονήσουμε γνωμοδότηση για την πρόταση σχετικά ε, με την ηλεκτρονική δημοσίευση της επίσημης εφημερίδας και κατόπιν μιλήσαμε για τις επόμενες επισκέψεις των αντιπροσωπιών της Επιτροπής μας και συζητήσαμε την επόμενη επίσκεψη στις 14 Ιουλίου. Απεβεβαιώσαμε την απόφασή μας για την επίσκεψη αυτή που είχε ήδη εγκριθεί από το Προεδρείο με κάποια όρια που δεν μας αρέσουν, αλλά αποφασίσαμε να δεκτούμε των αυτών. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στα θέματα που έχουμε να συζητήσουμε. Παρακαλώ, ο κύριος Γκερέριο. Ευχαριστώ πρόεδρε, καλημέρα σας. Δεν ξέρω αν καθυστέρησα και τις αναφέρετε αυτές τις πληροφορίες. Θέλω να ρωτήσω κάποια ομάδα ζήτησε η προθεσμία για τις τροπολογίες για την μεταρρύθμιση του άρθρου 70 να μετακινηθεί κατά μία εβδομάδα. Να έχουμε παράταση για μία εβδομάδα. Δεν υπάρχουν προβλήματα, λέει ο Πρόεδρος. Δεν το συζητήσαμε το θέμα αυτό, αλλά... Αν υπάρχει αίτημα από τον εισηγητή, μπορούμε να το πράξουμε. Ναι, δεν είναι δική μου η πρόταση. Νομίζω ότι υπήρχε μια πρόταση από το Λαϊκό Κόμμα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, και εγώ θα ήμουν υπέρ. Υπάρχει αυτή η πρόταση από το ΕΛΚ. Λοιπόν, επομένως θα έχουμε παράταση της προθεσμίας για την κατάθεση τροπολογιών κατά μία εβδομάδα. Να περάσουμε τώρα στο σημείο 9. Πρόκειται για την έκθεση Γκουαλτιέρη Τερκόφσκι αν θέλουν ε, να μας ενημερώσουν οι συνάδελφοι για αυτή την ε, έκθεση πρωτοβουλίας που είναι ιδιαίτερα σημαντική. Έχει ήδη Εμείς ε, ήδη διορίσαμε τους δύο συναδέλφους ως εισηγητές και ίσως μπορούν να μας δώσουν κάποιες πρώτες ενδείξεις για ποια μέθοδο σκοπεύουν να ακολουθήσουν για να προετοιμάσουν αυτή τη σημαντική έκθεση. Ο κ. Γκουαλτιέρη, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή είναι πολύπλοκη και νομίζω ότι απαιτεί και αρκετό χρόνο για την προετοιμασία της και κυρίως ε, πρέπει να έχουμε επαρκή χρόνο πριν από την εκπόνηση του πρώτου σχεδίου κειμένου γιατί πιστεύω ότι θα είναι σκόπιμο να μην περιοριστούμε στο προβληματισμό μας και στην έκθεση των ιδεών μας. Αντιθέτως, πρέπει να προσπαθήσουμε να συλλέξουμε ιδέες, να προβούμε σε ανάλυση, να συλλέξουμε προτάσεις από την πλευρά όχι μόνο των συναδέλφων, αλλά και από μια ευρύτερη κοινότητα την ακαδημαϊκή, την επιστημονική, την πολιτική και θεσμική κοινότητα και από την κοινωνία των πολιτών. Έτσι λοιπόν, πιστεύω ότι ως προς τη μεθοδολογία θα ήταν σκόπιμο να ακολουθήσουμε μια διαδρομή όπου θα εμπλακούν ε, διάφορα άτομα, δηλαδή ίσως να έχουμε και μια διαρθρωμένη εκρόαση εδώ φθινόπωρο. Ίσως και κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει πριν το καλοκαίρι και αναφέρομαι στο εξή ε, να καλέσει η ΑΦΚΟ κάποιες προσωπικότητες ε, τις οποίες καλό θα ήταν να ακούσουμε. Δεν θα μπω τώρα στην ουσία, διαφορετικά θα προβαίνω αντίφαση με όσα είπα πριν για τις προτάσεις ε, και τις ιδέες, αλλά να σας πω ποια είναι κατά την άποψή μου τα θέματα που πρέπει να εξετάσει η έκθεση αυτή. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από ένα αναλυτικό στοιχείο, από ένα στοιχείο ανάλυσης και αυτό είναι το εξή. Το γεγονός ότι αφενός ε, είχαμε μια πολύπλοκη μεταρρύθμιση με τη συνθήκη της Λισαβόνας, ε, η οποία έχει επίπτωση και στην πολυπλοκότητα της διαδικασίας μεταρρύθμισης των συνθήκων. Αυτό αφενός και φετέρου ήταν μια μεταρρύθμιση η οποία έχει τεθεί σε ισχύ εδώ και λίγο καιρό και η δυναμική αυτής της μεταρρύθμισης δεν έχει ακόμα πλήρως διερευνηθεί. Τώρα, από την άλλη, αμέσω μετά την ε, συνθήκη της Λισαβόνας, καταγράφηκαν κάποιες εξελίξεις ε, και κυρίως αναφέρομαι στον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης που οδήγησαν ε, τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιδράσει. Τώρα δεν μπαίνω στην ουσία για το αν απαντήσεις αυτές ήταν ή δεν ήταν κατάλληλες. Κατά την άποψή μου δεν ήταν, αλλά τέλος πάντων δεν είναι αυτό το ζήτημα. και αφενός να δείξουμε πώς μπορούμε να διευρύνουμε την ερμηνεία των συνδικών, παραδείγματος χάρη, ε, βάσει του άρθρου 122.2, το οποίο μας ε, απέτρεψε κατά κάποιο τρόπο ε, και το άρθρο 125 και από την άλλη μας οδήγησε να προσφύγουμε σε εξωτερικά μέσα πέρα των συνθήκων και αφενός ε, οι ίδιοι μηχανισμοί σταθεροποίησης ε, συνδέονται με τις συνθήκες αλλά έχουμε μια διακυβερνητική μορφή κυρίως του μηχανισμού χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και από την άλλη έχουμε και το Fiscal Compact, το Δημοσιονομικό, Σύμφωνο που είναι μια ε, συνθήκη διακυβερνητική. Και είδαμε ότι ίσως ε, προχωρήσαμε και ακόμη παραπέρα από όσα θα μπορούσε να έχει φανταστεί κανείς κατά την εκπόνηση της συνταγματικής ε, συνέλευσης και κατόπιν της συνθήκης της Αμόρας. Έχουμε λοιπόν μία διπλή διάσταση, μία διτή διάσταση. Έχουμε κάποια δυναμική που δεν έχει διερευνηθεί και έχουμε και κάποια καινούργια προβλήματα τα οποία δεν έχουν βρει στη συνθήκη την κατάλληλη απάντηση. Και εγώ νομίζω ότι πρέπει να προβληματιστούμε όχι όμως με έναν αφηρημένο τρόπο, με αφετηρία ε, έναν αφηρημένο τρόπο διακυβέρνησης, αλλά θα πρέπει να έχουμε σημείο αφετηρία στα προβλήματα που εκδηλώθηκαν και συγκεκριμένα το θέμα της ε, ε θεσμικής ασυμμετρίας, αν θέλετε, μέσα στις εισαγωγικά της Ευρωζώνης και των 27 και να αναλύσουμε και το είδος της απάντησης που δόθηκε, αλλά και τις δυνατότητες που προσφέρει η συνθήκη. Είτε σε ό,τι αφορά τη διεύρυνση των ε, νομοθετικών διαδικασιών, δηλαδή το πεδίο εφαρμογή ορισμένων ε, άρθρων 36, που κατά την άποψή μου δεν έχει διερευνηθεί ακόμα εις βάθος, Έχουμε βέβαια και το Τούπακ ε, και είναι πρώτοι κανονισμοί αυτή που βασίζονται στο 136. Κατά την άποψή μου το 136 θα μπορούσε να μας επιτρέψει να πάμε και παραπέρα. Είτε σε ό,τι αφορά συγκεκριμένε διαδικασίες όπως ενισχυμένε συνεργασίες, είτε σε ό,τι αφορά κάποια μέσα ενίσχυσης των αρμοδιοτήτων ε, της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω κατά νου τη ρήτρα της ευελιξίας. Έτσι λοιπόν, ε, αυτό το πεδίο εξέτασης ε, έχω κατά νου. Από την άλλη, θα πρέπει να ξεκινήσουμε να εξετάζουμε πιθανές ε, εξελίξεις, πώς θα μπορούσαν να εξελιχθούν οι συνθήκες σε σχέση με αυτά τα νέα προβλήματα που έχουν αναδυθεί. Και Πιστεύω ότι δεν πρέπει να περιοριστούμε στην ε, διάσταση της οικονομικής διακυβέρνησης, αλλά θα έπρεπε να αναλύσουμε και συναφή ζητήματα που αφορούν την ομιμότητα των ε, διαδικασιών λήψης αποφάσεων, δηλαδή τη δημοκρατική διάσταση, την ε, διοργανική ισορροπία και ε, ακριβώς την νομοθετική πρωτοβουλία του Προέδρου Συμβουλίου. Νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο ε, σε αυτές τις γενικές γραμμές θα πρέπει να κινηθεί η έκθεση, η οποία λόγω του πολύπλοκου χαρακτήρα της ε, και επειδή έχουμε και ισχυρή παρουσία μιας αναλυτικής διάστασης για τις ε, ουσιαστικές, τις υλικέ εξελίξεις που είδαμε μετά την έγκριση συνθήκη της Λισαβόνας, απαιτούν αυτή την ευρεία και μακρά διαδρομή και τη συμμετοχή διάφορων πρωταγωνιστών σε μια διαδικασία εκπόνησης του κειμένου. Και το κείμενο αυτό σίγουρα είναι πολύ πιο σημαντικό από τις δυνάμεις των ε, δύο ταπεινών εισηγητών. Ευχαριστώ κύριε Γκουαλτιέρη και τώρα θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Ταρκόφης και ο οποίος είναι σας. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Συμφωνώ προφανώς με όσα είπε ο Ρομπέρτο. Σας είχα πει νομίζω ότι με το που πήρα το πτυχίο μου το Πανεπιστήμιο Άρχισα να προετοιμάζω την ανάλυση από πλευρά Πολωνία τη ε, θεώρησή μα για τη συνθήκη του Άμστερνταμ. Και θυμάμαι ότι πριν τελειώσω καλά-καλά, ο καθηγητή μου μου είπε πρέπει να αρχίσει να αλλάζει τώρα ίσως ε, προσανατολισμό γιατί αλλάζει και η συνθήκη. Και δεν έχει νόημα να κοιτάξει πιο πολύ βάθος τα θεσμικά ζητήματα. Με την συνθήκη τη Λισαβόνας που παρακολουθήσαμε κάπως από το περιθώριο, γιατί δεν ξέρω αν θυμάστε, είχαμε λιγότερες ψήφους από την Ισπανία. Προσπαθήσαμε να επηρεάσουμε όμως εξελίξεις και με τον ε, Πρωθυπουργό Μπούζεκ. Είχαμε φτάσει και μέχρι την Νίκαια προσπαθώντας να πείσουμε για τα δικά μας επιχειρήματα. Και αφού πέρασα μερικές άϊπνες νύχτες, μου είπε ο καθηγητής μου πάλι Α, τώρα πρέπει να αλλάξει πάλι, διότι και η νίκαια θα τροποποιηθεί. Και χωρίς να θέλω να σας κουράζω με την ε, πανεπιστημιακή μουσιοδρομία. Είναι πολλέ οι φορές που έχουμε ακούσει ότι δεν πρόκειται να γίνουν άλλες αλλαγέ θεσμικέ, αλλά αποδεικνύεται ότι βρισκόμαστε ως προς τους θεσμούς σε μια διαρκή ροή και αυτό που κάνουμε εν προκειμένου με τον Ρομπέρτο είναι ότι προσπαθούμε να συλλέξουμε και να καταγράψουμε σε ένα έγγραφο τα θέματα, χωρίς βέβαια να φιλοδοξούμε να εκφράσουμε τις θέσεις του Κοινοβουλίου και να προκαταλάβουμε την προσοχή γύρω θεσμικών μεταρρυθμίσεων, αλλά προσπαθούμε να καταγράψουμε τα σημεία στα οποία χρειάζεται συζήτηση. Επομένως, τα καταγράφουμε, τα ταξινομούμε, τα αναλύουμε και το πιο σημαντικό νομίζω είναι, γιατί υπήρξε και μια φάση όπου όλοι υπερασπίζονταν τι συνθήκε Λισαβόνα λέγοντα ότι είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε περαιτέρω. Αλλά τώρα που κατά ο κουρνιαχτό είναι, πιστεύω, η ώρα να ρίξουμε μια ματιά συνθήκε Λισαβόνα, τι συνθήκε εφαρμογή τη, τη θεσμική τη ισορροπία, τι θεσμικέ τη ισορροπίε, τα επιτεύγματα, αν επιτύχαμε αυτά τα οποία επιδιώκαμε με τη διαπραγμάτευση. Και, εν πάση περιπτώσει, ποιο θα ήταν ο δρόμο πέραν αυτή. Άρα, μετά τη Λισαβόνα, μετά το δημοσιονομικό ε, σύμφωνο, πρέπει να αναλύσουμε την κατάσταση και κυρίως τον κίνδυνο κατακαιρματισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να κοιτάξουμε και τη μεταβλητή γεωμετρία και άλλα πιθανά σενάρια, όλα τα πιθανά σενάρια για το μέλλον. Καταγράφουμε λοιπόν όλες τις θέσεις που συζητήθηκαν εδώ τα τελευταία τρία χρόνια στην Επιτροπή των Σταγματικών Υποθέσεων. Υπογραμμίζουμε τα πιο σημαντικά ζητήματα που πιστεύουμε ότι θα πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη τη στιγμή που θα συζητηθούν θεσμικές αλλαγές. Και γι' αυτό πιστεύω ότι χρειάζεται και αυτή η περίοδος α, μελέτης αναλογισμού. Γι' αυτό και ξεκίνησα με την ομάδα αναλογισμού Westendorf του 2005. Βέβαια, εν προκειμένου θα ήθελα να πω ότι ελπίζω ότι θα έχουν καλύτερη μοίρα, ότι θα έχουμε καλύτερα, καλύτερη μοίρα από ότι εκείνη, γιατί η ομάδα αναλογισμού είχε υποθεί ότι ούτε η ομάδα ήταν ούτε αναλογισμό έκανε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ελπίζω ότι θα μπορέσουμε εμεί και σαν ομάδα να δράσουμε και κοινή θέση να διατυπώσουμε. Αυτό είναι ο στόχο για τον οποίο αγωνιζόμαστε, Ρομπέρτο και εγώ. Και επίση ελπίζουμε ότι θα συλλέξουμε και θα αναλύσουμε αρκετέ θέσει, αλλά πάνω απ' όλα ότι θα μπορέσουμε και να εξετάσουμε, ε, να συζητήσουμε, να μελετήσουμε τι θέλουμε για το μέλλον και ποιες είναι οι προτεραιότητες που ορίζουμε. Αλλά πάνω απ' όλα τώρα θα ήθελα να ακούσω τους συναδέλφους. Για σε αυτή τη σύντομη περίοδο αναλογισμού θα ήθελα να ακούσω τις δικές σας προτεραιότητες και τις δικές σας επόψεις για αυτή την έκθεση με το κάπως συμβιλικό όνομα. Τίτλο. Ευχαριστώ. Ήδη έχουν ζητήσει κάποιοι συνάδελφοι το λόγο. Καταρχήν, συνάδελφος Επτήμερ, σας παρακαλώ να είστε σύντομοι γιατί στις 10 θα ξεκινήσουμε και την ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Πριν από πολύ καιρό, όταν σπούδαζα αστυνομική, μου λεγόταν ότι μου είχε υποθεί ότι ο Ιουστιβιανός τον επεξεργαζόταν στι νεαρέ του, θεωρούσε ότι θα, ήταν, ε, ότι θα έμεναν στον αιώνα τον άπαντα ενισχύ. Και γι' αυτό νομίζω ότι είναι χρήσιμο να ξεκινάμε με αυτή την ε, τοποθέτηση, ότι δηλαδή υπάρχουν πάντα ανάγκε για τροποποίηση στην νομοθεσία. Αυτό φαντάζομαι ισχύει και για την τωρινή συζήτηση, για την νομοθεσία που θα συζητήσουμε και θα προετοιμάσουμε εδώ. Δεν υπάρχει δηλαδή τίποτε το οριστικό και μόνιμο. Οτιδήποτε πράξουμε, οτιδήποτε αναλύσουμε, θα πρέπει να το αναλύουμε έχοντα υπόψη ότι θα τροποποιηθεί αργότερα. Αυτά για να συμμετάσχω στη συζήτηση και για να πω ότι θα πρέπει και όσοι δεν ανέχουν στο Κοινοβούλιο να συμμετάσχουν στη διαδικασία αυτή με μια ακρόαση ενδεχομένω, Ρομπέρτο, με, με ένα μεγάλο συνέδριο στο οποίο θα μπορούσαν να συμμετάσχουν όχι όλοι διότι δεν είναι δυνατόν, αλλά όσο δυνατόν περισσότεροι ε, ενδιαφερόμενοι και εμπλεκόμενοι φορείς η Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια κάνουμε κάποιες διακρίσεις τις οποίες, τις οποίες δεν προβαίνουν όσοι βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά βλέπουμε ότι χάνει την νομοποίηση της η Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε μέρα και αναπτύσσεται ένα αίσθημα εχθρικό απόρριψης και γι' αυτό νομίζω ότι χρειάζεται νέα πνοή Πρέπει να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών και αυτό θα το καταφέρουμε με μια καλύτερη παρουσίαση των όσων πράττουμε. Πράγμα το οποίο ακόμα δεν έχουμε επιτύχει. Δεν περνάει δηλαδή το μήνυμα και νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον από την Ουγγαρία μπορώ να το διαβάσω αυτό και να πω ότι αυτό είναι και ο κύριο αγώνα τον οποίο αποδίωμε. είναι ένα θέμα το οποίο συζητούμε στην Επιτροπή μας από το 2004 τουλάχιστον που είμαι εγώ μέλος, αλλά εν πάση περιπτώσει βλέπουμε ότι δεν έχει επιληθεί ακόμη. Δύο ζητήματα πιστεύω θα πρέπει ιδιαιτέρως να καλυφθούν διαφορετικά σε ένα βαθμό. Το ένα είναι, θα έλεγα, η εποπτεία, η επιτήρηση των εξουσιών που εκχωρούνται τώρα, αλλά υπάρχει και το ευρύτερο ζήτημα, δηλαδή του τρόπου με τον οποίο να ασκείται από τις Βρυξέλλες η εξουσία, είτε πολιτική είτε δικαιική, νομική, και της ε, απόστασης την οποία αισθάνεται ο πολίτης από τα κέντρα αυτά εξουσίας. Γιατί ο πολίτης αισθάνεται αδύναμο σε σχέση με το κέντρο εξουσίας που είναι οι Βρυξέλλες και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό λοιπόν καλό θα ήταν να συστήσουμε τους μηχανισμούς που θα μπορούσαμε ενδεχομένως, να οικοδομήσουμε προκειμένου να αναπτύξουμε τον ε, σύνδεσμο με τον πολίτη. Να επανασυνδέσουμε τον πολίτη με την εξουσία. Όταν μιλούμε βέβαια για 500 εκατομμύρια πολίτες, προφανώς έχουμε να κάνουμε με κάτι το πολύ δύσκολο και το ε, καινοφανές. Ποτέ δεν έχει αναπτυχθεί αντίστοιχο εγχείρημα στο παρελθόν. Άρα ναι, ξέρουμε ότι δεν υπάρχει προηγούμενο παράδειγμα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να απευθύνουμε ένα μήνυμα αποτελεσματικά προ 500 πολίτε με τρόπο διαφορετικό από τι 10 εκατομμύρια ή 15 ή 18 εκατομμύρια πολίτε ή 80 εκατομμύρια που έχει μεγαλύτερη χώρα μέλο Ευρωπαϊκή Ένωση Γερμανία, από ό,τι θυμάμαι. Εν περιπτώσει, το θέμα δεν είναι μόνο η ποσότητα, γερμανια απο οτι θυμαμαι Με περιπτωσει το θεμα δεν ειναι μονο η ποσοτητα αλλα για να ε, παραφράσω λίγο τον Καρλ Μάρξ, ε, η ποσότητα μερικές φορές μετατρέπεται και σε ποιότητα. Εν ολίγης, θα πρέπει να έχουμε να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση ισχυρότερη παρουσία μέσα στα κράτη-μέλη, να συμμετέχει στο βαθμό του δυνατού στον δημόσιο διάλογο που αναπτύσσεται σε τοπικό επίπεδο. Δηλαδή να λέμε ότι ναι, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποιοι σε τοπικό σε εθνικό επίπεδο που δεν μεταφέρουν απαραίτητα τα μηνύματά του ή το, ε, τις απόψεις μέσω, ε, μέσω του Συμβουλίου, μέσω των κρατών μελών δηλαδή και ότι μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους σε επίπεδο κράτους μέλους εμπλεκόμενοι φορείς, δηλαδή ενδιαφερόμενοι φορείς που θα πρέπει να πλησιάσουμε. Αυτό είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να αναπτύξουμε τον ε, διάλογο Και μου ότι όσο πιο πολύ συζητούμε, τόσο πιο πολύ θα είναι και εκείνοι που θα αναγνωρίζουν εν τέλει τι πράττει η Ευρωπαϊκή Ένωση και που θα ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερο. Και έτσι το μήνυμα θα ε, μεταφέρεται ευχερέστερα. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει σε πολιτικούς όρους να επιχειρηματολογούμε. Δεν αρκεί να το πράττουμε αυτό μόνο σε νομικούς ή δικαιικούς μόνο όρους, όρους νομοθεσίας δηλαδή. Και επίσης, Ρομπέρτο, επισημαίνεις ότι είναι περίπλοκη όλο αυτό το εγχείρημα, αλλά ακριβώς γι' αυτό, αυτό πρέπει και να επισημάνουμε, να πούμε, να μιλήσουμε για τις περίπλοκες δομές. Δεν νομίζω ότι αρκεί δηλαδή με ένα φυλάδιο ή με ένα βιβλίο τύπου ε, οικονομική διακυβέρνηση για αρχαρίους να προσπαθήσουμε να καλύψουμε όλο αυτό το πλέγμα που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά ε, δεδομένου ότι μάλλον εμείς αντιλαμβανόμαστε καλύτερα από όλους τι είναι, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να απευθύνουμε, ε, να, στείλουμε την εξήγηση και το μήνυμα στο δυνατόν ευρύτερο κοινό. Ασφαλώς και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι σε θέση να αντιληφθούν το μήνυμα αυτό και απλώς θα πρέπει να τους αγνοήσουμε και να τους παραμελήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Γκερέρο. Ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή και τον Ρομπέρτο είναι τα δύο ρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Ρομπέρτο και ο Ραφάλ. Είναι μια διανοητική περιπέτεια αυτή στην οποία έχουμε μπει. Θα συνεισφέρω και εγώ λέγοντας ότι και το δικό μου το διδακτορικό είχε να κάνει με το κοινοβουλευτικό έλεγχο της κυβέρνησης. Και όταν ήρθα εδώ στο Κοινοβούλιο, είχα φανταστεί ότι θα μπορούσα να εφαρμόσω εδώ όλα αυτά τα οποία είχα ερευνήσει για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο των άλλων θεσμικών οργάνων. Βέβαια, περνώντας ο καιρός, είδα ότι ο έλεγχος εξαφανίζεται σιγά-σιγά όσο τα θεσμικά όργανα, ιδιαίτερα το Συμβούλιο, τα κράτη-μέλη, βρίσκουν μηχανισμούς για να αποφεύγουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να αποφεύγουν ακριβώς ε, αυτόν τον έλεγχο. Ε, αυτή είναι και η δικιά μου μικρή απογοήτευση. Είμαστε σε ένα παράδοξο όσον αφορά την εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας και το παράδοξο είναι ότι ό,τι νέο έφερε η συνθήκη της Λισαβόνας και είχε να κάνει με την θεσμική φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως τέτοιας, ε, αυτό είτε σταμάτησε, βλοκαρίστηκε, είτε έχασε την επικεντρωθήκαμε στην αντιμετώπιση της κρίσης με μηχανισμούς οι οποίοι δεν προβλέπονται από τη συνθήκη της Λισαβόνας ή δρούμε στο περιθώριο της συνθήκης της Λισαβόνας. Αυτή λοιπόν η έκθεση είναι μια σημαντική έκθεση γιατί ακριβώς λαμβάνει υπόψη αυτή την αντίφαση, την αντιφατική πραγματικότητα, αυτό το παράδοξο. Θα λέγω ότι είναι μια διαδικασία στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι, όχι μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλαδή. Γι' αυτό και πιστεύω ότι είναι καλή ιδέα να έχουμε επαφές, να προσκαλέσουμε εμπειρογνώμονες ε, από την κοινωνία των πολιτών επίσης, να έρθει εδώ κόσμος. Υπάρχουν δύο αρχές της πραγματικότητας που δεν πρέπει να ξεχνάμε και αναφέρθηκαν σε αυτές και ο Ρομπέρτο και ο Ραφαέλ. Η πρώτη αρχή είναι ότι η μεταρρύθμιση, μάλλον ο προβληματισμός μας, να το πω καλύτερα έτσι, επικεντρώνεται σε ειδικά ζητήματα. Δεν είναι δηλαδή ένας προβληματισμός για τη συνταγματικότητα, πώς ιδεοδός θα έπρεπε να είναι ή πώς θα μπορούσαμε σε έναν ιδανικό κόσμο να έχουμε μια θεσμική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι, κατεβαίνουμε στην πραγματικότητα, εντοπίζουμε συγκεκριμένα προβλήματα και από αυτά πια προσπαθούμε να λύσουμε. Η πραγματικότητα είναι, και όλοι οι συνταγματολόγοι, και έχουμε εδώ πολλούς το γνωρίζουν καλά, είναι η πραγματικότητα λοιπόν ότι οι μεταρρυθμίσεις ήθιστε να γίνονται κοιτώντας προς τα πίσω. Δηλαδή, κοιτάμε τι προβλήματα είχαμε στο παρελθόν για να λύσουμε προβλήματα του μέλλοντος. Συνεπώς, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι θα προτείνουμε ανάλογα με το τι αντιμετωπίσαμε στο παρελθόν, ναι, αλλά να μην περιοριστούμε μόνο στα προβλήματα του παρελθόντος, γιατί τότε η πρότασή μας δεν θα ανταποκρίνεται στα προβλήματα του μέλλοντος. Αυτή λοιπόν είναι μια αρχή της πραγματικότητας. Άρα ναι, με να κοιτάμε πίσω, με ανοιχτό πνεύμα, με φιλοδοξία, αλλά να βλέπουμε όχι μόνο τι θέλουμε να λύσουμε σήμερα, αλλά και το τι έχει γίνει στο παρελθόν. Να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή που θα μας βοηθήσει να λύσουμε τα προβλήματα του μέλλοντος. Βέβαια, το να μπορεί κανείς να προβλέψει το μέλλον δεν γίνεται. Θέλω να πω στον Ραφαέλ αυτό που είπε για την ομάδα προβληματισμού, ότι στην Ισπανία υπάρχει ένα όργανο που είναι το Ανώτατο Συμβούλιο Επιστημονικών Ερευνών. Και ο διευθυντής του είπε κάποια φορά ότι έχω την εντύπωση ότι κανένα από αυτά τα τέσσερα πράγματα δεν είναι ούτε συμβούλιο, ούτε ανώτατο, ούτε ερευνητικό, ούτε επιστημονικό. Αυτά. Ευχαριστώ. Εδώ βλέπω ότι συνεισφέρετε όλοι ε, με τις ακαδημαϊκές σας ε, σπουδές, ε, με τις διπλωματικές εργασίες, τη διδακτορικά σας κτλ. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Νταφ. Ευχαριστώ κι εγώ για όλα αυτά. Με τη σειρά μου και η ομάδα μου θα ήθελε να αναφερθεί σε αυτή την έκθεση για την διαφοροποίηση στην διακυβέρνηση και να πει ότι θα ήθελε να είναι υπεράνω της διακυβέρνησης ακριβώς. Γιατί δεν είμαστε εμεί που φτιάχνουμε την ατζέντα για τη διακυβερνητική του 2015. Ελπίζω λοιπόν πριν από το τέλος αυτής της εντολής ως Επιτροπή, παρόλα αυτά, να ετοιμάσουμε μία έκθεση η οποία θα έχει σαν αποτέλεσμα η ατζέντα να εμβαθύνει ακόμα περισσότερο. δεν θα πρέπει να είναι απλώς και μόνο πώς θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των ε, κρατών ε, και του εκλογικού σώματος που δεν ακολουθεί την ομοσπονδιακή οδό. που θέλει πλειοψηφία. Βέβαια το πρόσχημα είναι και από πού ξεκινάει η έκθεση αυτή για τη διαφοροποιημένη διακυβέρνηση. Είναι μια απόφαση που λήφθη τον Δεκέμβριο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να αντιμετωπίσει τη Βρετανική στάση που ήταν να αρνηθεί ο Πρωθυπουργό ε, Κάμερον και να βάλει βέτο στην αλλαγή της ε, συνθήκης και να μην ισχύσει αυτή και για τους 27. Όμως η προοπτική να μπορέσουμε να μεταρρυθμίσουμε τις συνθήκες και με τους 27 συν την Κροατία. Σταματάει εδώ, τελειώνει. Νομίζω ότι η Λισαβόνα ήταν η τελευταία συνθήκη η οποία δεσμεύει όλες τις χώρες μέλη υπέρ ε, των ίδιων πολιτικών στόχων και τους δεσμεύει σε μία και την ίδια νομική τάξη. Αν θέλουμε λοιπόν το επόμενο στάδιο να έχει κάποιο νόημα, το επόμενο στάδιο δηλαδή συνταγματικών εξελίξεων, πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό της διαφοροποίησης ή της απόκλησης. Η διάσωση του ευρώ απαιτεί μία δημοσιονομική ένωση και μία ομόσπαδη οικονομική διακυβέρνηση. Γνωρίζουμε όμως ότι δεν θα συμπεριληφθούν εκεί όλα τα κράτη-μέλη. Νομίζω λοιπόν ότι οι εισηγητές έχουν την τάση να είναι πιο φιλοσοφικοί και να διευρύνουν τη συζήτηση αυτή για την φύση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Καλό θα ήταν να μείνουν στην ε, μία και μεγάλη πρόκληση και αυτό θα πρέπει να είναι και το καθήκον τους. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, γι' αυτό θα δώσω το λόγο στον αδελφό Σαντερκέτ και κατόπιν ε, δεν θα σας δώσω το λόγο για να απαντήσετε. Θα μπορέσετε να λάβετε υπόψη όσα υπόθηκαν ε, για την επόμενη παρουσίαση του εγγράφου σας. Παρακαλώ, κύριε Σαντερκέτ. Øh, øh, Ευχαριστώ τους συζητητές για την παρουσίασή τους. Ο τίτλος του κειμένου έχει να κάνει με τη διαφοροποίηση στην διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα σχετικά συνταγματικά προβλήματα. Θα ήταν καλό λοιπόν να έχουμε μία ιδέα για το τι θέλουμε να κάνουμε αναλύοντας ε, τα προβλήματα αυτά. Ποιος είναι ο στόχος μας, σε τι βαθμό θέλουμε να προχωρήσουμε σε λύσεις. Νομίζω ότι εδώ υπάρχει μια μεγάλη διαφορά στην προσέγγιση. Ανάλογα με το σημείο κίνησης του καθενός. Ο σχεδιασμός λύσεων είναι κάτι πολύ σημαντικό είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν λύσεις. Πρέπει να αποφύγουμε να έχουμε ένα κατάλογο επιτροπών κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή το θέμα δεν είναι να φτιάξουμε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο με επιθυμίες, το να θέλουμε να συμπεριληφθούν ε, λύσεις στη συνθήκη μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, αυτό μπορεί να είναι μια επιθυμία. Το FSF είναι μηχανισμός που θα κρατήσει βέβαια κάποια χρόνια. Ακόμα και αν ε, συμπεριληφθούν στη συνθήκη ή όχι. Πρέπει λοιπόν να είμαστε ρεαλιστές όσον αφορά τη σημερινή κατάσταση. Δεν μπορεί δηλαδή να αρκούμεθα σε κατάλογο επιθυμιών. Πριν από μερικές ε, μέρες στην Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού είχαμε μια ακρόαση για το δημοκρατικό και κοινοβουλευτικό έλεγχο των διάφορων μηχανισμών ε, σταθερότητων του EMS, ε, του EFSF και το ελεγκτικό συνέδριο, μηχανισμό σταθεροποίησης δηλαδή κλπ, είπε ότι ε, έπρεπε να οργανώσει μια συνάντηση με τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια και το έκανε. Για να εμπλακούν ακριβώς τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια και έτσι να μπορέσει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο να λειτουργήσει. Το πρόβλημα που έχουμε εδώ είναι ότι το εθνικό επίπεδο τελικά παίζει πιο σημαντικό ρόλο Ακριβώς γιατί υπήρξε η διακυβερνητική συμφωνία. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, συνεπώς, στα πλαίσια της διοργανικής συμφωνίας. Μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές λύσεις. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι να λάβουμε υπόψη μας και αυτόν τον προβληματισμό, αυτή τη διάσταση. Χάρη σε ακροάσεις πιστεύω ότι μπορούν να συμμετάσχουν και άλλοι φορείς στην όλη διαδικασία. Λοιπόν, ε, είπα ότι δεν θα δώσω το λόγο για απάντηση, αλλά είδα τον κύριο Γκερέρο ότι ζήτησε το λόγο και θα σημειώσουν οι συγητές όσα υπόνονται. 30 δευτερόλεπτα ήθελα να υπογραμμίσω κάτι που είπε ο κύριος Γκουαλτιέρη ότι πρέπει να διερευνήσουμε τις δυνατότητες που μας προσφέρει η σημερινή δομή. Αυτό ήταν πρόβλημα το προηγούμενο 1,5 χρόνο Οπότε είχαμε διαφορετική αντίληψη στο Κοινοβούλιο σχετικά με την αναγκαιότητα εισαγωγή μεταρρυθμίσεων ή όχι και τη δυνατότητα να πετύχουμε του ίδιου στόχου ε, χρησιμοποιώντα με κατάλληλο τρόπο το εφιστάμενο πλαίσιο. Αυτή τη συζήτηση την κάναμε σε σχέση με το Δημοσιονομικό Σύμφωνο και νομίζω ότι πρέπει να υπογραμμιστεί αυτό το θέμα, έτσι όπως είπε και ο Ρομπέρτο, να χρησιμοποιήσουμε αυτά που έχουμε σήμερα στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Ευχαριστώ. Έτσι λοιπόν συζητήθηκε το θέμα σε γενικές γραμμές και οι συγκριτές μας έχουν τώρα το καθήκον ε, να λάβουν όλα αυτά υπόψη και μας ανέφεραν και μια μεθαλλική ένδειξη για τις μελλοντικές εργασίες. Θα περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερική διάταξης, το σημείο 6, προπολογισμός 2013, εντολή για τον τριμερή διάλογο. Ο κύριος Γκερέρο είναι ο εισηγητές. Θα θυμάστε ότι στην προηγούμενη συνεδρίαση ακούσαμε τον εισηγητή για το γενικό προπολογισμό, τον κύριο Λαβία, και εδώ ε, έχουμε να κάνουμε με το θέμα της διαδικασίας προπολογισμού που ισχύει από τη Συνδίκη της Λισαβόνας για να προετοιμαστεί η πραγματική πρόταση προπολογισμού της Κομισιόν και θα δούμε τι ενδείξεις μπορούμε να έχουμε για την τριμερή διάλογο. Κύριος Γκερέρο, ευχαριστώ πολύ. Από την πλευρά μου θα είμαι σχετικά σύντομος, ε, καθώς ένα ουσιαστικό μέρος που σχετίζεται με τη γνωμοδότηση αυτή έχει να κάνει με τα συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία που υπάρχουν ήδη στην πρόταση της Κομισιόν για τον προπολογισμό του 2013 και αυτά τα αριθμητικά στοιχεία μόλις παρουσιάστηκαν χθες από την Επιτροπή και ε, θα αναφερθώ σε κάποια από αυτά συνοπτικά αλλά ε, και άλλα μέλη της Επιτροπής ε, φαντάζομαι ότι δεν έχουν ακόμη πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία, δεν τα γνωρίζουν, έτσι λοιπόν θα είναι δύσκολο να ανταλλάξουμε απόψεις για το θέμα αυτό. Όμως, εγώ θέλω να επισημάνω το εξής. Όπως γνωρίζουν ε, τα μέλη της Επιτροπής, εμείς πρέπει να διατυπώσουμε μία γνωμοδότηση για τον προϋπολογισμό που θα συμπεριληφθεί στις γνωμοδοτήσεις των διάφορων επιτροπών, έτσι ώστε η Επιτροπή Προϋπολογισμών να ε, προβεί στις διαπραγματεύσεις στον τριμερή διάλογο για τον προπολογισμό του 2013. Το χρονοδιάγραμμα που έχουμε είναι το εξή. Σήμερα παρουσιάζω αυτή τη γνωμοδότηση. Φυσικά θα ακούσω τι απόψει ε, που θα διατυπωθούν σχετικά με το θέμα αυτό. Θα υπάρχει προθεσμία για τι τροπολογίε ε, περί τα τέλη Μαΐου για να ψηφίσουμε και κατόπιν ε, να συμπεριλάβουμε το κείμενό μας στην πρόταση της Επιτροπής Προπολογισμών. Στη συνέχεια θα υπάρχει ένα δεύτερο έγγραφο για τα αριθμητικά στοιχεία, για τα συγκεκριμένα ποσά και σε μια διαδικασία που θα καθοριστεί από την Γραμματεία, την Προεδρία και τους συντονιστές θα πρέπει να εγκρίνουμε πριν από το καλοκαίρι ε, το κείμενο αυτό έτσι ώστε μετά το καλοκαίρι να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Η γενική ιδέα βάσει της οποίας συνέταξα το σχέδιο γραμμοδότησης είναι η εξής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί ενώπιον του μέλλοντος να ε, στρέφεται μόνο στη δημοσιονομική σταθερότητα, αλλά θα πρέπει να σκέφτεται και πώς θα βγει από την κρίση με μια ικανότητα οικονομικής παρέμβασης για μεγαλύτερη ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας από τη σημερινή. Όταν ε, συνεδριάσαμε με τον κύριο Λαβία, που είναι ο Γενικός Εισηγητής για τις διαπραγματεύσεις για τον προπολογισμό, Ε, παρήρχαν, μάλλον να πω ότι υπάρχουν και κάποια μέλη τη Επιτροπή Αφρικού που ίσω δεν συμφωνούν με τη θέση αυτή, που όμω νομίζω ότι βρίσκει σύμφωνη την πλειοψηφία, δηλαδή να προσδώσουμε περισσότερου πόρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να απαντήσει πιο κατάλληλα στην κρίση και για να υπάρξει μια όθηση στη δημιουργία θέσεων απασχόληση ε, και στην ανάπτυξη. Όμω από την ποσοτική σκοπιά αυτό δεν είναι ένα θέμα ιδιαίτερα σημαντικό για αυτή την Επιτροπή. Γιατί εμείς δεν είμαστε μια επιτροπή που ειδικώ εμπλέκεται σε μεγάλες επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά στο συγκεκριμένο ζήτημα, δηλαδή ως προς την εμπλοκή της συμμετοχής ΑΦΚΟ, έχει συμπεριληφθεί μια σειρά τυχόν πιο συγκεκριμένο στο κείμενο, όπως παραδείγματος χάρη, ότι το επόμενο έτος είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Ιθαγένειας και επίσης ε, το ότι τίθεται σε πρακτική εφαρμογή η νομοθετική πρωτοβουλία ε, των πολιτών η πιθανότητα να είναι αυτός ο τελευταίος προϋπολογισμός που θα εγκρίνουμε πριν από τις επόμενες ευρωεκλογές και Επομένως, πρέπει να έχουμε κατά νου αυτή την, την ε, εκλογική διαδικασία, με συγχωρείτε, κάτι που σημαίνει υποστήριξη και στα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, προκειμένου σε όλη την επικράτεια της Ένωσης ε, να ε, μπορέσουν να ενεργοποιήσουν ένα προβληματισμό των πολιτών επί των πολιτικών της Ένωσης. Αυτά είναι τα σημεία επί των οποίων ε, η γνωμοδότηση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων ε, θα πρέπει να αναφέρεται πιο συγκεκριμένα. Σύμφωνα με τα αριθμητικά στοιχεία που αρχικώς μας έδωσε η Κομισιόν, παρουσιάζοντας τον προπολογισμό, παραδείγματος χάρη, ενώ χάρη το κονδύλι Europe for Citizens, Ευρώπη για τους πολίτες, ε, διατηρείται στο ίδιο επίπεδο με πέρσι. Υπάρχει κάποια μείωση μάλιστα. Και για το Ευρωπαϊκό Έτος ε, των Πολιτών του 2013 υπάρχει μείωση εκεί σε σχέση με τον προπολογισμό που είχαμε το 2012. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί με κάποιο τρόπο, δηλαδή το επόμενο έτος ήδη θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή ο προπολογισμό που είχαμε το 12 και σε ό,τι αφορά στην ηλεκτρονική επικοινωνία υπάρχει κάποια αύξηση των κονδυλίων, όμως τα γενικά αριθμητικά στοιχεία του 2013 είναι παρόμοια σε μεγάλο βαθμό με τα νούμερα που είχαμε το 2012. Και επομένως δεν θα επιμείνουμε τώρα στα αριθμητικά στοιχεία γιατί θα υπάρχει δυνατότητα γι' αυτό. Αλλά εγώ ζητώ από τους συναδέλφους, από τα μέλη της Επιτροπής, αν είναι δυνατόν να συμφωνήσουν μαζί μου σε σχέση με τη γενική ιδέα ότι ο προπολογισμό της Ένωσης θα πρέπει να συνεισφέρει για την έξοδο από την κρίση και για τη γενική ιδέα ότι το καθήκον αυτή τη Επιτροπή είναι να αναφερθεί στην πρωτοβουλία των πολιτών, στο Ευρωπαϊκό Έτο των Πολιτών, στην επικοινωνία με του πολίτε και στη χρηματοδότηση στο πλαίσιο τη προεκλογική εκστρατεία για το 2014 και να έχουν κατά νου ότι η Κομισιόν να παρουσίασε ουσιαστικά τα ίδια κονδύλια πάνω κάτω που υπήρχαν το 2012, του ίδιους πόρους που είχαμε το 2012 και ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε όλα αυτά λεπτομερέστερα στο μέλλον. Πρόεδρος. Παρακαλώ. Κύριο Σόντεργκας. Όχι. Κύριε Ε, ε, ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πολύ σύντομα. Δεν μπορούμε να δώσουμε ποσά ακόμη και συγκεκριμένο προπολογισμό. Αλλά πάντως ευχαριστώ θερμά τον συγκεκριμένο κύριο Γκερέρου. Για, την, ε, για το κείμενο αυτό τη σύντομη αυτή γνωμοδότηση, πολύ καλή όμως. Νομίζω ότι πολύ σωστά επισημαίνει ότι πρέπει πια να μιλάμε όχι για περικοπές, αλλά για τομείς τους οποίους μπορούμε και πρόκειται να αυξήσουμε ή να ενισχύσουμε τον προπολογισμό. Μην ξεχνάμε ότι το 2013 θα είναι έτος που προηγείται ε, χρονιά εκλογών και θα είναι και έτος των Ευρωπαίων πολιτών. Επομένως πρέπει να δώσουμε έμφαση σε αυτή τη διάσταση. Χρειάζεται περισσότερη χρηματοδότηση και χρειάζεται η χρηματοδότηση να είναι ε, στο ύψος των περιστάσεων, να αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. λοιπόν, άλλε ερωτήσει. Βλέπω θέλετε να προσθέσετε κάτι, κύριε Γκέρερο. Όχι, κατόπιν όσο είπε ο κύριο Αντάργα. το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να αναγνωρίσω ότι αυτό ήταν συγητή ε, πέρσι και κατά κάποιο βαθμό εμπνεύστηκα από το έργο του. Σα ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Πολύ ωραία. Ολοκληρώνουμε λοιπόν και το σημείο αυτό και να περάσουμε στις προφορίες. Έχουμε ορισμένες εκθέσεις να ψηφίσουμε. Καταρχήν την έκθεση γκουρμάει. Έτσι λοιπόν, θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Έχουμε τέσσερις τροπολογίες συμβαστικές που έχουν παρουσιαστεί όπως γνωρίζετε. Και θα ψηφίσουμε την πρώτη. Λοιπόν, πρέπει να περάσουμε στις πληροφορίες. Χθες, ε, επειδή υπήρξε ανάγκη να δώσουμε κατευθείαν ε, το λόγο στην Αντιπρόεδρο τη Επιτροπή, ε, εγώ ξέχασα να σας πω ότι έπρεπε να εγκρίνουμε τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης. Έτσι λοιπόν, ε, θέλω να σας ε, ρωτήσω αν συμφωνείτε να εγκριθούν τα πρακτικά. Ξέχασα να σας ρωτήσω χτες, δεν βλέπω αντιρρήσεις. Έτσι λοιπόν, ε, θεωρείτε ότι εγκρίνονται τα πρακτικά κατά τα λοιπά. Έχετε λάβει τα έγγραφα ήδη. Τώρα, αν δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση, μπορούμε να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία και θα ψηφίσουμε τις συμβαστικές ε, τροπολογίες και την συμβαστική τροπολογία D, δέλτα. Ποιος είναι υπέρ, παρακαλώ, τα. Κατά. Τρεις ψήφοι κατά. Αποχές. Μία αποχή. Εγκρίνεται.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 Ποιος είναι υπέρ, παρακαλώ. Άνατας χειρός. Κατά. Αποχές. Μια αποχή. Εγκρίνεται. Μπορούμε τώρα λοιπόν να ψηφίσουμε το chair of the. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Τέσσερις ψηφικά κατά αποχές. Μία αποχή. Και προχωράμε. Αφήνουμε αυτή την ψηφορία κατά θα περάσουμε στο σημείο 3. Νομίζω ότι αφορά εδώ την παράγραφο 1, χωρίς τους όρους members μέχρι το issue of. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ψηφίζουμε τώρα για τις λέξεις αυτές. Πρώτα τις αποκλείσαμε. Ποιος είναι υπέρ λοιπόν. Κατά. Τρεις. Αποχές. Ένας. Λοιπόν, και τώρα έχουμε την εκπροστή ψηφοφορία για την παράγραφο 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Μία αποχή, τέσσερις ψήφοι κατά. Και τώρα θα ψηφίσουμε για την παράγραφο 6, υπέρ. Κατά. Έτσι λοιπόν καταπίπτουν όλες ε, οι τροπολογίε υπόλοιπε και θα περάσουμε στην τροπολογία 2. Υπέρ. Για την τροπολογία 2. Παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Στη συνέχεια... Πρέπει να πάμε στην τροπολογία 27. Μόνο το τμήμα που αφορά τα εδάφια 3 και 4, γιατί τα υπόλοιπα ε, προφέρθηκαν από την ε, ψηφοφορία που είχαμε πριν. Έτσι λοιπόν να ψηφίσουμε τώρα μέσα στα όρια αυτά την τροπολογία 27. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. Να πάμε τώρα σε συμβαστική τροπολογία α. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και περνάμε στη συμβαστική τροπολογία β. Β. Υπέρ. Κατά. Τρεις. Αποχές. Ένα. εγκρίνεται. Περνάμε στη τελευταία συμβιβαστική τροπολογία, Σι, γάμα, υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Φτάνουμε στη τελευταία ψηφορία για την παραγραφό 5, τροπολογία 9, DAF, υπέρ. Κατά. Εποχές. Εγκρίνεται. Συγγνώμη, απορρίπτεται, απορρίπτεται. Ναι, απορρίπτεται, απορρίπτεται. Και περνάμε στην τελική ψηφοφορία για το κείμενο που στροποποιήθηκε υπέρ. Κατά. Μία ψήφος κατά. Αποχές. Τρεις, τέσσερις. Εγκρίνεται λοιπόν. Το σχέδιο ε, είχαμε 17 ψήφους υπέρ, 4 αποχές και μία ψήφο κατά. Μπορούμε λοιπόν τώρα να προχωρήσουμε στην επόμενη έκθεση. Ο κύριος Νταφ. Πρόεδρε, θα ήθελα να παρακαλέσω να γίνει μια ονομαστική ψηφοφορία στο σημείο αυτό. Επικαλούμενο στο 195.3 του κανονισμού. Gaddaf vuole anticipare quella che sarà la sua, la sua proposta di... Μάλιστα, από ό,τι βλέπω θέλετε εδώ να προτρέξετε σε σχέση με την ε, γενική πρότασή σα. Ε, πάντοτε θέλω όσα κηρύττω να τα θέτω σε εφαρμογή, Πρόεδρε. Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, υποστηρίζετε από τους συναδέλφου η πρόταση αυτή. Δεν βλέπω την υποστήριξη. Ποιος είναι υπέρ. Ποιο είναι υπέρ στην πρόταση αυτή. Λοιπόν, να προχωρήσουμε με ονομαστική ψηφοφορία. Τι πρέπει να κάνουμε με τεχνική σκοπιά. Κύριε Νταφ, αυτή η πτυχία Μήπως εσείς θέλετε να μας καθοδηγήσετε, να μας πείτε για να την ονομαστική ψηφοφορία την επιθυμείτε μόνο για την τελική ψηφοφορία ή το ζητάτε και για τις επιμέρους ψηφοφορίες. Εκτός μικροφώνου τα σχόλια. Η ουσιαστική τροπολογία είναι υπαριθμόν 3. Και για την τελική ψηφοφορία. Θα ήθελα κάτι τέτοιο. Βέβαια, αν δεν ε, εγκριθεί η υπαριθμό 3, τότε η ουσία όλης της έκθεσης αλλοιώνεται. Είναι καινογράμμα. Δηλαδή, δεν θα είχε νόημα να προχωρήσουμε πέραν της τροπολογίας 3. Σε σχέση τον κύριο Βίλα. Προτείνουμε να προτείνω να καταψηφίσουμε την τροπολογία του. Αλλά να δούμε τι θα γίνει με την τροπολογία 3, αν θα εγκριθεί ή όχι. Λοιπόν, απαντάτε εσείς λοιπόν, θέλετε ηλεκτρονική ψηφορία για την τροπολογία 3. Τα υπόλοιπα δεν σας ενδιαφέρουν, έτσι είναι. Κύριε Σταφ. πιθανόν και για την τελική ψηφοφορία. Αλλά ας δούμε πρώτα τι θα γίνει με την τροπολογιατρία. Πολύ ωραία. Α, μάλιστα, δεν έχετε κάρτα. Και Τζαρκόφσκι. Ναι, ε, έχετε όλη την κάρτα. Τι γίνεται κύριε Τσαρκόφσκι, δεν έχετε κάρτα. Να σας ε, καλέσω λοιπόν τον καθένα ξεχωριστά. Να ψηφίσουμε λοιπόν ηλεκτρονικά και να καλέσουμε ονομαστικά όσοι δεν έχουν κάρτες. Έτσι λοιπόν όσοι δεν έχετε κάρτες θα κληθείτε να τοποθετηθείτε ουσιαστικά, να ψηφίσετε ουσιαστικά. Λοιπόν, ψηφίζουμε την τροπολογία 3 του εισηγητή. Άρχεται η ψηφορία. Ε, ε, ε Ψηφίσατε όλοι. Μάλιστα. Κύριε Ταρκόφσκι, ψηφίσατε κατά. Κύριε Χαβινέρ, υπέρ. Λοιπόν, έχετε την κάρτα μάλιστα. Για να δούμε πέρα τη ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Ναι, βλέπουμε το αποτέλεσμα. 6 υπέρ και 12 κατά. Συγγνώμη, συγγνώμη, πρέπει να προσθέσουμε και τους συναδέλφους που δεν είχαν κάρτα. 13 κατά λοιπόν και 8 υπέρ. Απορρίπτεται λοιπόν. Εγώ παρακαλώ να καταγραφεί ότι καταψήφισα, δεν δουλεύει η κάρτα μου. Την έχω μαζί μου όμως. Λοιπόν, είναι σε σαφή τα πράγματα. Βλέπουμε στην ηλεκτρονική μορφή 12 κατά 7 υπέρ. Έχω προσθέσει μία ψήφο υπέρ και μία κατά και έλαβα υπόψη και τη δήλωση του κ. Ταρκόφης και Χέρνερ. Τώρα ο κ. Λεβενή λέει ότι καταψηφίζει γιατί δεν λειτουργήσε η κάρτα του. Αυτό σημαίνει ότι. 9 υπέρ και 13 κατά. Συγγνώμη. Συγγνώμη. καταψήφισε ο συνάδελφος, όχι δεν υπερψήφισε. Διορθώνω. Διορθώνω τον εαυτό μου. 8 υπέρ, 14 ψήφοι κατά. Λοιπόν, εντάξει, δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, πολύ ωραία. Να περάσουμε τώρα στην τροπολογία 1 που αποσύρεται. Δεν θα το ψηφίσουμε λοιπόν καθόλου. Και η 3 αποσύρθηκε. Έτσι λοιπόν μας μένει μόνο η τροπολογία 2. Παρακαλώ υπέρ. Chi è Κατά. Απορρίπτεται, είναι προφανές. Ε, ε, ε, Κύριε Πρόεδρε, προφανώς έχει εξουδετερωθεί πλέον αυτή η έκθεση. Δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε τώρα, ούτε σε τελική ψηφοφορία. Δεν υπάρχει τίποτε να ψηφίσουμε δηλαδή. Μάλιστα, σας ευχαριστώ κύριε Νταφ. Έτσι έχουν τα πράγματα. Εγώ κανένα δεν ήθελα να δολοφονήσω, απλώς όμως ε, δημοκρατικά καταγράφω την ψήφο. Θα έπρεπε τώρα λοιπόν να εξετάσουμε το κείμενο που αφορά την ερμηνεία του άρθρου 117 του κανονισμού. Εγώ είμαι εισηγητής, όπως ξέρετε για το θέμα αυτό. sono La Burma e le chiede da un attimo la parola per una questione rispetto a ieri. C'è la mozione d'ordine o comunque una richiesta di parola. Non abbiamo etima από την κυρία Γκουρμάη, θέλει να πάρει το λόγο. Λοιπόν, πριν να πάμε σε αυτό το τελευταίο σημείο, στη 13 της ημερησία διάταξη, να δώσω το λόγο στην κυρία Γκουρμάη. Ε, Ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα αυτή την ευκαιρία, μια και είναι όλοι εδώ παρόντες, σχεδόν μέλη τη Επιτροπή. να αναφερθώ σε, μία από τις, ε, σε ένα από τα θέματα που ε, διατύπωσα χθε προ την κυρία Ρέντινγκ, που έκανε μια πάρα πολύ καλή παρουσία όπως συνήθως εχθές, αλλά τα νέα εκατομμύρια ευρώ τα, τα περσινά, από τα οποία 2,8 δαπανήθηκαν για το Euronews, γιατί στη συνέχεια ε, γιατί είχε ματαιωθεί το εγχείρημα για, την πανευρωπαϊκή τηλεοπτική δικτύωση, το πανευρωπαϊκό τηλεοπτικό δίκτυο και ήθελα να ρωτήσω τι έγιναν τα υπόλοιπα χρήματα μετά τα 2,8 έως τα 9 εκατομμύρια, τι έγινε. Θα ήθελα λοιπόν η Επιτροπή, σας, η Επιτροπή μας να με στηρίξει στο αίτημα να απευθύνουμε μια γραπτή ερώτηση προς την κυρία Ρέντινγκ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν τα χρήματα αυτά, δεν ξέρω αν έχουν εξαφανιστεί, αλλά είναι πολύ σημαντικό ποσό και πρέπει να είμαστε ενήμεροι. Εάν έχει απο... δαπανίσει για τα κονδύλια αυτά η κυρία Ρέντινγκ, πρέπει να ενημερωθεί το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Chairman, I think, uh, Πρόεδρε, η κυρία Γκούρμαϊ νομίζω έχει πολύ εύστοχα επισημάνει ότι πρέπει να επιμείνουμε η Επιτροπή να απαντήσει. Ε, προτείνω λοιπόν η Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή να υποστηρίξει το αίτημα. Μάλιστα. Υποστηρίζουμε λοιπόν την πρόταση της κυρία Γκουρμάη. Να περάσουμε τώρα. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Να περάσουμε στο σημείο 13 που αφορά την ερμηνεία του 17, όπως ξέρετε κατόπιν ετοίματος της υπόθεσης εξωτερικών της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων Κοιτάξτε, ε, το έχουμε ξανασυζητήσει το θέμα. Είναι απλό το ζήτημα. Επί της ουσίας, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων μας ζητά να τοποθετηθούμε ή μερμηνία, ή με του κανονισμού επί του θέματος σύμφωνα με το οποίο αν ε, η Επιτροπή και το Συμβούλιο δεν απαντήσουν μέσα σε 7 εβδομάδες σε κάποιο ερώτημα ενό Ευρωβουλευτή θα πρέπει το θέμα να μπει στην ημερήσια διάταξη της Αρμόδιας Επιτροπής ε, στην πρώτη συνεδρίαση πριν να λήξει προθεσμία. Έτσι λοιπόν ε, δηλώνω την ησυχία της Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ε, γιατί ε, φοβάται ότι ε, θα ήταν, γινόταν πάρα πολύ βαριά η μερισία διάταξη και ενώ θα έπρεπε να εξεταστούν άλλα σημαντικά θέματα, θα ε, παρέμβαιναν αυτές οι ερωτήσεις. Ε, εγώ δεν νομίζω ότι πρέπει να τροποποιήσουμε κάτι, αλλά απλώς να προσπαθήσουμε να κάνουμε τα πράγματα με το σωστό τρόπο. Δηλαδή, όχι απλώς να έχουμε μόνο κατά νου το άρθρο 117, το άρθρο 117 λέει στην πρώτη σύνοδο της Αρμόδιας Επιτροπής τίθεται στη για διάταξη το ζήτημα για το οποίο δεν απάντησαν Κομισιόν και Συμβούλιο. Αυτό δεν μπορούμε να το κυρώσουμε, αλλά υπάρχει ακριβώς και το άρθρο 193 του κανονισμού που προβλέπει ο πρόεδρος της Επιτροπής ε, είναι αυτός που θα καταρτήσει τη μεσία διάταξη, όχι μόνο δηλαδή τη μεσία διάταξη εξαρτημητική σειρά 1, 2, 3, 4, αλλά στη δική του διακριτική ευχαίρεια θα είναι να καθορίσει ποια στιγμή μπορεί να συζητηθεί το θέμα που έχει τεθεί στη μεσία διάταξη της πρώτης συνεδρίασης και από την άλλη η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει την μεσία διάταξη του συνολό τη. έτσι λοιπόν μπορεί να ζητήσει την αναστολή, την ε, διαγραφή κτλ. Γι' αυτό προβλέπει βλέπετε ευελιξία και κατά την άποψή μου νομίζω ότι πρέπει να κατευθυνθούμε ως εξή, να αντιμετωπίσουμε τον κανονισμό έτσι ώστε να αποφύγουμε ε, αυτή την ε, δυσκερή κατάσταση την οποία φοβάται η Επιτροπή ΑΦΚΟ. Έτσι λοιπόν ε, νομίζω ότι αν είναι δυνατόν και συμφωνείτε να ψηφίσουμε και σήμερα. Αλλά νομίζω ο κύριος Γκουλατιέρη θέλει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υποθέτω ότι δεν είναι ένα ζωτικό ζήτημα. Εγώ, όπως ήδη έχω πει, έχω μια τεχνική ως αμφιβολία σε σχέση με το πόσο βάσιμες είναι οι ερμηνείες αυτές. Προσωπικά, πιστεύω ότι ίσως ε, θα έπρεπε να διαγράψουμε το να βάλουμε στην μισή για την επόμενη συνάντηση και να λέμε ότι πρέπει απλώς να είναι στην μισή διάταξη. Καθώς δεν πρόκειται για ένα ξεκαθαρό ζήτημα, θα θέλω να ακούσω και τη γνώμη των συναδέλφων. Και αυτό το θέμα είναι να αφηθεί μεγαλύτερη ευκαιρία για το πότε θα συζητηθεί το θέμα. Έτσι λοιπόν, μειώνεται η πίεση που ασκείται στην Επιτροπή. Εγώ νομίζω ότι είναι ένα πραγματικό πρόβλημα και με αυτόν τον τρόπο θα λυνόταν με ένα πιο διαφορετικό τρόπο παρά με το να μπει στην ημερική διάταξη και κατόπιν να αποφασίζεται να αφαιρεθεί αμέσως μετά. Όμως, ε, καθώς μιλάμε για ένα θέμα που δεν είναι και τόσο σημαντικό. Δεν θέλω να κατέβω και στα χαρακόμματα και να υπερασπίσω έντονα την άποψή μου. Απλώ ε, το καταθέτω εδώ για να τοποθετηθούν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι από την Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Γκολτιέρη. Σας ευχαριστούμε για το επικοδομητικό σας ε, πνεύμα και το πνεύμα συνεργασίας. Ο κύριος Μάρτιν. Ευχαριστώ. Στηρίζω την επιστολή σας η Επιτροπή Εξωτερικών ε, Υποθέσεων αντιδράει στο ότι υπάρχει στην ημερήσια διάταξη. Είναι για προσπληροφόρηση. Πρόκειται για ερωτήσεις προς απάντηση. Δεν πρέπει να υποθέσουμε ότι θα συζητηθεί δύο-τρεις ώρες η κάθε ερώτηση. Εγώ προσωπικά θα ήμουν υπέρ γιατί πιστεύω ότι πιέζει τα άλλα θεσμικά όργανα προκειμένου να συμμορφωθούν προς το άρθρο 117 δεν πρέπει να αντιδρούμε σε αυτά που λέει το άρθρο 117. Πιέζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντάει πιο γρήγορα στα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κύριε Σέφνερ, Πρόεδρε, ευχαριστώ και εγώ πολύ σύντομα. Καταρχάς ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε την ε, νοοτροπία άλλων ε, κοινοβουλευτικών επιτροπών. Πρέπει απλά να δίνουμε ερμηνείες ή προτάσεις ερμηνείας. Εγώ προσωπικό συμφωνώ με τη δική σας. Και δεύτερον, θα ήθελα να επισημάνω ότι είναι απαραίτητο να δίνουμε ερμηνεία για διευκρίνηση και όχι να προσπαθούμε πάντα να κάνουμε τροποποίηση στον κανονισμό. Εάν διαγράψουμε την φράση όμως next meeting, προσεχή συνεδρίαση, τότε παραμένει μάλλον ασαφές το πότε θα γίνει αυτό και νομίζω ότι θα πρέπει καταρχήν να ισχύει ότι η συζήτηση θα γίνεται στην προσεχή συνεδρίαση. Με την ερμηνεία όμως μπορούμε να έχουμε ένα περιθώριο ε, χειρισμών ευρύτερο, το οποίο ισχύει για ολόκληρη την Επιτροπή και αν χρειαστεί μπορεί να γίνει ψηφοφορία. Εγώ νομίζω ότι είναι καλύτερο λοιπόν να δώσουμε ερμηνεία για να διευκρινιστεί η υπόθεση και να ε, εκφράσω, θα ήθελα να εκφράσω τη συμφωνία μου στην ερμηνεία αυτή. Λοιπόν, καθώς ε, ο κύριος ε, Γκουαλτιέρη έδειξε πνεύμα συνεργασίας, θα μπορούσαμε να υιοθετήσουμε αυτή την πρόταση ερμηνείας. Ποιος είναι υπέρ, παρακαλώ, ένα τεσχύρος. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Ευχαριστούμε. Έχουμε ομοφωνή έγκριση και περνάμε στο επόμενο σημείο που αφορά τις εξεταστικές επιτροπές. Αρκετά σημαντικό το θέμα αυτό και θα δώσω το, μάλλον και η συγκεκριτή είναι ο κ. Μάρτιν. Εμεί όμω στην πραγματικότητα έχουμε ήδη ψηφίσει τον έγγραφο του κ. Μάρτιν, αλλά δεν είχε μπει ακόμα στην υπηρεσία διάταξη τη Ολομέλεια, ε, γιατί υπάρχουν ε, κάποιε αμφιβολίε μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Έτσι λοιπόν ο κύριος Μάρτιν ε, ανέλαβε να διερευνήσει το θέμα, να δει αν μπορεί να βρει μια λύση για να πάμε στην ψήφο στην Λομέλεια. Κύριε Μάρτιν, έχετε το λόγο για να μας πείτε αν είναι δυνατό κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δίκιο έχετε. Οχτώ μήνες τώρα βρίσκεται σε κρεμότητα αυτό το θέμα από τον Οκτώβριο. Το έχουμε συζητήσει στην Επιτροπή μας και δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να το βάλουμε στην Ολομέλεια. Ελπίζω με τη στήριξη των άλλων πολιτικών ομάδων να συμπεριληφθεί στην Ολομέλεια του Μαΐου τη δεύτερη. Να σα θυμίσω, οι περισσότεροι θα το θυμόσαστε, ποιο είναι το ιστορικό υπόβαθρο. Με τη συνθήκη της Λισαβόνας ε, προθούνται οι ρυθμίσεις όσον αφορά την ε, δημιουργία εξεταστικής επί των πραγμάτων επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα θυμόσαστε ότι όταν είχαμε την Εξεταστική Επιτροπή εκούι, δεν είχε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επαρκές αρμοδιότητες ώστε να μπορεί να ζητάει έγγραφα ή να επιβάλλει την κλήτευση μαρτύρων ή να επιβάλλει την εκπόνηση υπομνημάτων κτλ. Γι' αυτό λοιπόν θέλαμε μια ισχυρή εντολή. Θεωρούσαμε ότι ήταν ισχυρή, αλλά δεν μπορούσαμε να παρεκκλίνουμε από αυτήν βέβαια ποτέ. Οι σκιώδεις συζητητές συνεργάστηκαν και με τα άλλα θεσμικά όργανα και η Γραμματεία, την οποία και θέλω να ευχαριστήσω για την βοήθειά τη στις τεχνικές συζητήσεις που είχαμε κυρίω με το Συμβούλιο. Αυτό που προσπαθώ εγώ να κάνω εδώ είναι να διαπραγματευτώ με την Προεδρία τη Δανία και να καταλήξουμε σε συμβιβαστικέ θέσει. Πρέπει να σας πω ότι η Προεδρία της Δανίας ήταν ιδιαίτερα συνεργάσιμη. Όταν πρώτο συζητήθηκε στο Συμβούλιο το θέμα, η αντίδραση του Συμβουλίου ήταν αρνητική. Πρέπει να σας πω ότι θα το είχαν απορρίψει. Όμως οι Δανείοι προσπάθησαν να συζητήσουν με διάφορα μέλη του Συμβουλίου και να εξηγήσουν τη λογική που βρίσκεται πίσω από τη δικιά μας τη στάση. Ο Επίτροπος Εύκοβιτς επίσης ήταν ιδιαίτερα συνεργάσιμος και βοήθησε να περάσουν διάφορες τροπολογίες. Έτσι κατέληξα και εγώ σε διαβούλευση, αλλά όχι απαραίτητα και σε συμφωνία με όλους τους σκιώδεις, ε, κατέληξα σε κάποιες τροπολογίες. Οι σκιώδεις ίσως να μην συμφωνούν με όλες, Πάντως, εγώ πρότεινα να υποβληθούν ε, στην Ολομέλεια όλες αυτές οι τροπολογίες και εφόσον ε, συμφωνήσουν είπε ο κύριο Βίλαν, δεν θέλω εδώ τώρα βέβαια εγώ να μιλήσω για τον κύριο Βίλαν, αλλά ξέρω ότι είναι πάρα πολύ επιφυλακτικό προκειμένου να ε, συμφωνήσουμε να συμφωνήσει με τις τροπολογίες. Αλλά υπάρχει και ο Άντριου, εδώ και ο ελπίζω να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Οι τροπολογίε αυτές δεν θα ικανοποιήσουν όλους εδώ στην Επιτροπή μας. Ούτε και σημαίνει ότι αυτόματα θα αντισδεχτούν τα άλλα θεσμικά όργανα. Πάντως ο λόγος που τις προτείνω είναι πρώτα απ' όλα ότι τα άλλα θεσμικά όργανα ε, σκέφτονται ότι α, έτσι και περάσει την έκθεσή του το κοινοβούλιο, τελείωσε. Δεν είναι σωστό. Έτσι κι αλλιώς πρόκειται για μια νέα, αν όχι και μοναδική διαδικασία που είναι το κοινοβούλιο που κάνει πρόταση και τα άλλα δύο θεσμικά όργανα πρέπει να τη δεχτούν και ιδιαίτερα η Κομισιόν αισθάνθηκε ότι έτσι και περάσει από την Ολομέλεια το κείμενο αυτό δεν θα μπορεί να υπάρξει καμία τροποποίηση. Δεν είναι αλήθεια αυτό, γιατί μετά η ρύθμιση θα πάει στη διαπραγμάτευση. Πάντως πριν μπούμε στον τριμερή διάλογο, καλό θα ήταν το Κοινοβούλιο να δείξει ότι είναι διατεθειμένο με ευελιξία να προσεγγίσει τις άλλες θέσεις των άλλων δηλαδή θεσμικών οργάνων. Και αυτό προσπάθησα και να κάνω. Γι' αυτό είναι τόσο ήπια η δικιά μου η προσέγγιση. Πρέπει να ξέρετε ότι ιδιαίτερα το Συμβούλιο θεώρησε ότι είναι υπερβολικά νομικίστικη η διατύπωσή μα. Ότι δηλαδή θέλουμε οι εξεταστικές αυτέ επιτροπέ να μοιάζουν πάρα πολύ με δικαστήρια. Δεν είναι έτσι. Θα σας δώσω κάποια παραδείγματα που θα μπορούσα να μετακινηθώ. Άρθρο 11 για παράδειγμα. Εδώ έχουμε αλλάξει όχι βέβαια την ουσία, αλλά την διατύπωση για να το δεχτεί το Συμβούλιο. Δηλαδή, δεν μιλάμε απαραίτητα για μαρτυρίες, αλλά λέμε για ε, υπομνήματα υπαλλήλων. Στο άρθρο 15 επίσης κρατάω τον τίτλο που είναι «Μάρτυρες», αλλά αντί να μιλάω για μάρτυρες και τα λοιπά, μιλάω για άτομα στη συνέχεια. Εννοείται ότι έρχονται να καταθέσουν, αλλά μιλάω για άτομα και, για άτομα και όχι για μάρτυρες και όχι για μαρτυρίες, μήπως αυτό βοηθήσει το Συμβούλιο. Αλλάζει γλώσσα δηλαδή, οπότε ίσως να φανεί στο Συμβούλιο λιγότερο νομικιστικό. Κάτι πιο ουσιαστικό είναι το ότι τα άλλα θεσμικά όργανα ανησυχούν για το κατά πόσο κυκλισμένο το θυρών θα γίνονται οι μαρτυρίες. Και τώρα εγώ θέλω να εμείνω στην ουσία, αλλά ότι τα στοιχεία έτσι κι αλλιώς θα τα ακούσουμε και πριν. Δηλαδή όταν έρθει κάποιος και κλεισμένο το θυρών να καταθέσει, πρώτα θα ακούσουμε τους λόγους για τους οποίους κλητεύεται το άτομο αυτό και μετά θα δούμε ε, για την μαρτυρία του και το θυρών. Να, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα το δικαίωμα κλήτευσης. Άρθρο 17. Εδώ ξέρω ότι ορισμένοι συνάδελφοι πιστεύουν ότι το παρακάνουν. Κοιτάξτε, ακούστηκαν πολλές ανοησίες για το άρθρο 17. Και ο κύριος Άγνιου δεν είναι εδώ, τέλος είναι ε, υπεύθυνος μιας ε, ομάδας επικεφαλής ε, λέει ότι τι είναι η βασίλισσα εδώ, η επιτροπή αυτή, η οποία θα υποχρεώνει τον κόσμο να έρχεται. Νομίζω ότι φαίνεται από το άρθρο αυτό ότι δεν το βλέπουμε έτσι. Εμείς πιστεύουμε ότι εμείς μπορούμε να ζητήσουμε από διερμηνείς να έρθουν και να παρευρεθούν στην ε, κάθε μαρτυρία. Τίποτα άλλο. Κατέληξα λοιπόν σε ένα συμβιβασμό που λέει ότι η Επιτροπή, τα κράτη-μέλη είτε συμμορφώνονται είτε εξηγούν γιατί δεν συμμορφώνονται. Είτε συμμορφώνονται δηλαδή με το αίτημά μας ή κάποιος αξιωματούχο, υψηλαιστάμενος ή ένα επίτροπο έρχεται και εξηγεί γιατί ο συγκεκριμένο υπάλληλο δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην κλήτευση που γίνεται. Μπορεί να μην είναι ιδανικό, αλλά στην κατάσταση που βρισκόμαστε πιστεύω ότι είναι η καλύτερη λύση. Και άλλε αλλαγέ. Ευχαριστώ να συζητήσω μαζί σα εφόσον θέλετε. Πάντως, στόχος μας είναι να δείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι να μετακινηθούμε για να πλησιάσουμε τι θέσει των άλλων θεσμικών οργάνων και παραμένουν βέβαια κάποια θέματα προς διαπραγμάτευση. Κάποιοι μπορεί να έχουν διαφορετικές κόκκινες γραμμές. Εγώ έχω μία. Και αυτή είναι ότι πρέπει να γίνεται ποιοτική βελτίωση της κατάστασης. Αν έχουμε και καταλήξουμε σε ένα πακέτο μέτρων που βελτιώνουν την κατάσταση, εγώ θα είμαι ικανοποιημένο. Δεν είμαι διατεθειμένο να κολλήσω στο ένα ή στο άλλο ζητηματάκι. Το θέμα είναι να προχωρήσουμε προ βελτίωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μάρτιν. Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το έργο. Κύριο Ντάφ. Ε... Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δουλειά του. Είναι σημαντικό, πιστεύω, να αντιληφθούμε πόσο ιδιαίτερη φύση έχει αυτό το εγχείρημα είναι το δεύτερο θέμα, όπως προβλέπει η συνθήκη με το δικαίωμα πρωτοβουλία. Και δεδομένου ότι δεν έχουμε καταφέρει μεγάλη πρόοδο στην άλλη διαδικασία που έχουμε πρωτοβουλία, μπορούμε νομίζω να ε, επιδιώξουμε εδώ τουλάχιστον να διεκδικήσουμε μια πιο ισχυρή παρουσία. Και είναι πολύ σημαντικό και λεπτό το θέμα. διότι έχει να κάνει και με το εθνικό δίκαιο, όπου οι όροι που ισχύουν ε, ανακράτος μέλο για τη λειτουργία των εξεταστικών επιτροπών ε, μπορούν να επικύλουν σημαντικά από κράτος μέλος σε κράτος μέλο. Οι εξεταστικές επιτροπές σε ορισμένα κράτη μπορεί να έχουν πολύ συχνή παρουσία, έως μόνιμη, σε άλλα όμως σχεδόν μηδενική. Άρα θα πρέπει με κάποιο τρόπο να βρούμε μια συμφωνία μεταξύ μας, αλλά και με το Συμβούλιο για το θέμα αυτό. Επίσης, Συμφωνώ με την πρόταση να καταφύγουμε στην Ολομέλεια για να εγκρίνει αυτές τις ε, τροπολογίες και εκ μέρους της Άλντε, τη θα τις εγκρίνουμε. Αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε να επιληφθούν πλήρως οι ομάδες μας αυτών των θεμάτων, να τα συζητήσουν προσηκόντως για να δούμε τα θέματα. Σας διαβεβαιώ ωστόσο ότι θα υπάρξουν πολλές, ε, ε, πολλοί διχασμοί και στο εσωτερικό των ομάδων, όπως άλλωστε και στο θέμα των διαδικασιών για τις εκλογές. Όπως είπα λοιπόν, δεν μπορώ να δεσμευθώ σε ε, σχέση με το τελικό αποτέλεσμα, αλλά το τελικό συμπέρασμα, αλλά σας διαβεβαιώ ότι θα το υπογράψω για την Ολομέλεια. Κυρίω το θέμα των ενδεκών βοηθημάτων. έτσι ώστε να μην ακροτεριαστεί τελείως η Εξεταστική Επιτροπή ως διαδικασία. Γιατί θα κληθούμε να δώσουμε και απαντήσεις ως προς την αξιοπιστία τουλάχιστον ορισμένων περιστάσεων της διαδικασίας όχι πάντοτε, αλλά εάν φτάσουμε μέχρι τον τριμερή διάλογο που θα φτάσουμε, θα ήθελα να επισημάνω ότι θα θίξω το ζήτημα, ή σκοπεύω να θίξω το ζήτημα των ενδίκων βοηθημάτων κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης. Ευχαριστούμε κύριε Νταφ. κύριος Βίλαντ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μάρτιν έκανε μια πολύ δεξιδική παρουσίαση. Είναι γνωστό νομίζω ότι σε ένα σημείο έχω κάποιες επιφυλάξεις. Έχουμε συμφωνήσει ωστόσο με τους συναδέλφους από το ΕΛΚ ότι θα δεχθούμε την πρόταση αυτή, αλλά όπως είπε ο κύριος δεν θα πρέπει να το ακροτηριάσουμε το πακέτο αυτό με τις προτάσεις. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει και σε επίπεδο Συμβουλίου. Και θα ήθελα να αναφερθώ σε, μια, σε ένα έργο λογοτεχνικό γερμανικό που έχουμε το, την εικόνα ενός γίγαντα, υποτίθεται, ο οποίος όμως από μακριά φαίνεται να τεράστιος, αλλά στην πραγματικότητα είναι μόνο μια σκιά. Αυτό λοιπόν είναι το μήνυμα που θέλω να στείλω, ότι δεν πρέπει αυτό το νομοθέτημα να μετατραπεί σε έναν ε, σκιώδη γίγαντα, χωρίς δηλαδή σάρκα και οστά. Οι προτάσεις είναι σημαντικές, μπορεί να έχουν και σημαντικό πολιτικό αντίκτυπο και πιστεύω ότι θα πρέπει ο μάρτυρας ή όποιος είναι να μην είναι σε θέση του μόνος του να αποφασίσει εάν θα, ζητήσει, εάν θα δώσει μαρτυρία ε, και των θυρών. Θα πρέπει να είναι σε θέση να εξηγήσει τους λόγους γιατί ζητεί την απόρριτη αυτή διαδικασία, έστω σε μια συνεδρίαση και κλεισμένων Και πάντως Εάν αποφασιστεί ότι δεν είναι ικανοποιητικό αυτό το αίτημα, τότε μπορεί και να ε, δοθεί η, να ληφθεί η απόφαση ότι επιτρέπεται στο μάρτυρα να μην ε, παραστεί στο, στην Εξεταστική Επιτροπή. Αλλά και πάλι πρέπει να υπάρχει αιτιολόγηση. Το επόμενο όμως λογικό βήμα είναι το εξής, ότι εκείνος ο οποίος θα έρθει να δώσει μαρτυρία θα πρέπει να είναι δεσμευμένος, να είναι υποχρεωμένος να δώσει αληθινή μαρτυρία, να μιλήσει ειλικρινά. Και γι' αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί από τα κράτη-μέλη και να δεσμευτούν τα κράτη-μέλη ότι η ψευδορκία σε περίπτωση ε, μαρτύρα ενό πληρωματή τη Επιτροπή Εξεταστική θα πρέπει να ε, βαρύνεται με τι ίδιε κυρώσει με αυτέ που ισχύουν για μια αντίστοιχη εθνική διαδικασία. Είπε όμω και ο κύριο Ντάφ ότι δεν υπάρχουν πάντοτε αυτέ οι διαδικασίε και αυτή η νοοτροπία σε όλα τα κράτη-μέλη και γι' αυτό και το ζήτημα τη ποινική ευθύνη είναι πολύ σημαντικό. Ε, το ζήτημα της, ε, ψήφου, της μειοψηφίας πρέπει νομίζω να υπάρξει, πρέπει να καταγραφεί αυτή, ε, δεχομένως ενισχυμένη μειοψηφία, για τη μορφή της ενισχυμένης μειοψηφίας στην Επιτροπή. Μετά, Σε άλλα ουσιαστικά ζητήματα δεν έχουμε τοποθετηθεί ακόμα ρητά. Περιμένουμε μια πιο επιφυλακτική στάση. Αλλά δεν θέλω να αναφερθώ στην εντύπωση που ενδεχομένως θα δινόταν σε σχέση με τις συμφωνίες πρώτης ανάγνωσης που ακούστηκαν και νωρίτερα ότι ίσως ε, να, δοθεί εντύπωση ότι προσπαθούμε με την ε, νομοθεσία αυτή να πιέσουμε για το ζήτημα της πρώτης ανάγνωσης. Γι' αυτό λοιπόν καλό θα ήταν και ο ε, εισηγητής μας με τους σκιώδεις εισηγητές να παρουσιάσουν το κείμενο σαν ενιαίο έργο, σαν κοινό έργο που το υποστηρίζουν όλοι, ώστε να μην δοθεί η εντύπωση ότι υπάρχουν κάπου ρογμέ στον τοίχο σε αυτό που μπορεί να παρουσιάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά ότι είναι γρανιτένιο πραγματικά. Ευχαριστώ πολύ, κύριο Σέφνερ. Ευχαριστώ. Έτσι μια σειρά από ζητήματα ουσίας. Εγώ πάντως θα ήθελα προς το παρόν αν και είναι πολλά αυτά που θα είχα να πω, να μην αναφερθώ στην ουσία, αλλά στη διαδικασία. Και θα ήθελα να πω σαφώς ότι δεν είμαι βέβαιος πως είναι ευφιές το προσευχές βήμα όπως περιεγράφει. Εδώ μιλούμε για μέσω άσκησης ε, του δικαιώματος ε, του ελέγχου ή της εξέτασης, όπως λέγεται στη συνθήκη της Λισαβόνας, του δικαιώματος που έχει αναγνωριστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που εξυπηρετεί τα συμφέροντα του πολίτη. Έτσι λοιπόν, ε, μπορούμε να ελέγχουμε και την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Και είναι προφανές ότι δεν ενθουσιάζονται η Επιτροπή και το Συμβούλιο στην προοπτική να χορηγηθεί αυτό το εργαλείο στα χέρια του Κοινοβουλίου. Έχω συζητήσει με τον κύριο Μάρτιν και με μία μόνο ψήφο είδαμε ότι υιοθετήθηκε η νομική βάση, η, βάση μάλλον, η βάση των γράφων, μια πολύ καλή βάση, ξέρουμε ότι δεν μπορούν να λυθούν τα πάντα, αλλά είναι πολύ σημαντικό να καταγραφεί ότι το Κοινοβούλιο θεωρεί πολύ σημαντικό και ότι είναι αυτή η βάση για τη διαπραγμάτευσή μας. Θεωρώ ότι δεν θα κερδίσουμε σε κάθε σημείο από αυτά που επιδιώκουμε. Ούτως ή άλλως λέει, θα πρέπει να γίνει μια στάθμιση, μια ψηφοφορία στη συνέχεια για κάποιες ενδεχόμενες τροπολογίες και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να γίνει τριμερής ε, η διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Καλό θα είναι να μην κάνουμε διαπραγματεύσεις στο περιθώριο, ε, ή να προσπαθήσουμε μόνο να δούμε σε σχέση με τη δανική προεδρία τι θα μπορούσαμε να κερδίσουμε. Όχι, πρέπει να δούμε ξεκάθαρα η Επιτροπή και ολόκληρο το Συμβούλιο τι θέση έχουν και ποια είναι η κατάσταση ως προς την αντιπαράθεση, διότι δεν είναι πολύ σαφές ε, και δεδομένο πάντοτε το Συμβούλιο και, το, και η Επιτροπή θα είναι στο πλευρό μας και θα προσπαθήσουν να υποστηρίξουν τα δικά μας συμφέροντα, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις οποίες μπορεί η Επιτροπή να συμμαχίσει μαζί μας κατά του Συμβουλίου και του Μπαλίνου. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να έχουμε τυπικό τριμερή διάλογο, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πρέπει να φτιάξουμε, πιστεύω, μια ομάδα διαπραγματευτική και βέβαια τον είπε φθηνό του τον επικεφαλής της, αλλά πάντως να στηρίζεται η ομάδα αυτή από όλες τις πολιτικές ομάδες. Η πρόταση για τροποποίηση της έκθεσης ε, πριν την υποβολή της στην Ολομέλεια Δεδομένου ότι θεωρώ ότι ούτω ή άλλω θα πρέπει να γίνει τροποποίηση κάποια στιγμή, να γίνουν τροπολογίε δηλαδή στην έκθεση και μετά να κατατεθεί στην Ολομέλεια. Ε, η, η πρόταση λοιπόν αυτή να πάμε τώρα στην Ολομέλεια, σε πρώτη φάση, με προβληματίζει ω προ το τι εικόνα θα δώσουμε και βέβαια μην ξεχνάμε ότι μπορεί εδώ να συζητάμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ε, κοινοβουλευτική μα Επιτροπή, αλλά δεν είμαστε μόνοι μα. Είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο, παρόντε, μπορούν να παρακολουθήσουν τι λέμε. Επομένω, ε, Προφανώς ε, πρέπει να δώσουμε το μήνυμα ότι είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε, αλλά εντολή βάση για τη λήψη απόφασης του Κοινοβουλίου είναι αυτή την οποία από κοινού συμφωνήσαμε εδώ. Το να προτείνουμε εδώ τροπολογίες τόσο νωρίς ε, θα μπορεί να αποτελέσει ένα ε, μια πρώτα συμβασμού την οποία μόνο αργότερα θα μπορούσα εγώ να δεχθώ. Την ώρα που θα έρθει η ώρα δηλαδή για τις διαπραγματεύσεις. Γι' αυτό δεν πιστεύω ότι θα πρέπει τυπικά να ψηφίσουμε για τις τροπολογίες αυτές τώρα. Θα πρέπει να τις αφήσουμε ως πιθανές τροποποιήσεις του κειμένου Άλλωστε και με τον εισηγητή και τους πιο συγητές νομίζω τους έχουμε συζητήσει. Το να πάμε όμως τώρα στην Ολομέλεια, να απευθυνθούμε τώρα στην Ολομέλεια για να ζητήσουμε τροποποίηση της εντολής δεν είναι για μένα καλό μήνυμα. Είναι μάλλον μήνυμα αδυναμίας παρά μήνυμα ισχύω από πλευρά μας. Ω δείγμα δε συνεργασία, διάθεση για συνεργασία δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητο. Μόνο αποδυναμώνει τη θέση του Κοινοβουλίου κύριος Μπρόντς έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω αντίρρηση να κλητεύει ε, αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κυρίως ε, το Κοινοβούλιο. Αντιθέτως μάλλον μου αρέσει η ιδέα αυτή, αλλά για ε, προσώπους των κρατών μελών, αξιωματούχους των κρατών μελών, δεν νομίζω ότι είναι καλή ιδέα να τους υπαγάγουμε στον έλεγχο των ευρωπαϊκών οργάνων που ξέρετε ότι εγώ δεν συμπαθώ ιδιαίτερα αντίθετα με εσάς. Πάντως για τους ε, υπαλλήλου, ξέρετε ότι μια κυβέρνηση μπορεί να αρνηθεί την ε, παρουσία και την κλήτευση και μαρτυρία ενώπιον μια εξεταστική επιτροπής ε, μια κυβέρνηση για κάποιου λόγου. Ωστόσο εδώ βλέπω στην παράγραφο 17 ενώ ότι τα θεσμικά όργανα και ή σώματα ή ε, κράτη-μέλη ορίζουν τους ε, υπαλλήλου ή αξιωματούχους της κυβερνήσεως κτλ. Άρα δηλαδή μπορούν να αποφασίσουν αυτά τα ευρωπαϊκά όργανα. Και στο 17.3 επίσης αναφέρεται ότι μπορεί η Επιτροπή Εξεταστική να κλητεύσει συγκεκριμένο υπάλληλο ή μέλο του λοιπού προσωπικού κράτου μέλου για να καταθέσει σχετικά με θέμα το οποίο έρχεται των επαγγελματικών του υποχρεώσεων, εάν κρίνει κτλ. Αυτό λοιπόν ε, που ήθελα να επισημάνω είναι και γιατί ανησυχώ για τον ε, υπάλληλο, τον δημόσιο υπάλληλο. Ο υπουργό, το μέλο τη κυβέρνηση μπορεί όπω και να έχει να αντιδράσει, να αντισταθεί, έχει μια κάποια προστασία και εν περιπτώσει είναι ενήλικα. Ο δημόσιο υπάλληλο ενό κράτου λοιπόν όμω, ενό κρατικού μηχανισμού είναι υποχρεωμένο να τηρεί πάντοτε ουδέτερη στάση. Εάν κληθεί να δώσει μαρτυρία για το τι είδου συμβουλή έδωσε σε υπουργό σε μια συγκεκριμένη υπόθεση, μπορεί να δοθεί εντύπωση ότι αμφισβητεί τη ουδετερότητά του. Ή σε άλλη περίπτωση, αν του ζητηθεί να δώσει άποψη για αποφάσει που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο μια ε, κυβερνητική ε, διαδικασία, μπορεί η αποκάλυψη αυτών των πληροφοριών να τον θέσει ε, σε, στη θέση του κατηγορουμένου σε εσωτερικέ διαδικασίε, γιατί αποκαλύπτει επί παραδείγματι απόρριτε πληροφορίε. Ή, εν πάση περιπτώσει, θα ήθελε ο δημόσιο υπάλληλο να βρεθεί σε, ενώπιον διλήμματο να ε, δώσει αληθή μαρτυρία για ένα ζήτημα, ενώ ο Υπουργό ε, στέλνει μήνυμα διακριτικά ότι ίσω να μην είναι τόσο ειλικρινή ο δημόσιο υπάλληλο όσο μπορεί να απαιτείται να είναι ενώπιον τη επιτροπή αυτή. και γι' αυτό βρίσκεται ενώπιον ενό αφόρητου διλήμματο ε, ο ε, υπάλληλο. Λοιπόν, αν ε, δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσει, κύριε Μάρτιν, να ακούσουμε την αντίδρασή σα και την πρότασή σα για το τι θα κάνουμε. Για το τελευταίο σημείο. Όσο είπε ο συνάδελφος, έχει δίκιο για τα όσα είπε και γι' αυτό προτείνω στην τροπολογία στο άρθρο 7 παράγραφος 2 την ε, δυνατότητα τα κράτη-μέλη να αρνηθούν ε, να διορίσουν ε, κάποιο υπάλληλο να καθορίσουν κάποιο υπάλληλο, αλλά αν καθοριστεί κάποιο ε, υπάλληλο, όπω είπε ο συνάδελφο, ε, τότε έχουμε το δικαίωμα να του ζητήσουμε να πει την αλήθεια και να είναι ανοιχτό απέναντι στην Επιτροπή, αν το επιτρέπεται από το κράτο μέλο. Ένας άλλο ε, λόγος που μπορεί να φανταστώ ένα κράτο μέλο να μην επιτρέψει στον υπάλληλο να παρευρεθεί είναι επειδή παραδείγματο χάρη μπορεί να καλύπτεται από τι μυστικέ υπηρεσίε ή λειτουργεί δυνάμει εντολή του, Υπουργού. Όμως πρέπει να παρουσιαστεί ε, στην Επιτροπή και να εξηγήσει γιατί δεν είναι αυτό το κατάλληλο άτομο να παρουσιαστεί. Σας ευχαριστώ ε, για το όσα είπατε. Κύριε Βιλάν. δεν συμφωνώ 100% αλλά... Ε, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συμβαστική πρόταση. Ευχαριστώ τον κύριο Άννου που ε, θα υποστηρίξει κάποιες τροπολογίες που δεν τον ικανοποιούν απόλυτα και φυσικά αυτό θα σημαίνει ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε και θα βοηθήσει πάρα πολύ αν τουλάχιστον τρεις μεγάλες ομάδες προσυπογράψουν τις τροπολογίες. Κατανοώ τα τόσο είπε ο κύριος Χάφνερ και ειλικρινά και εγώ από εκεί ξεκίνησα. Και η δική μου άποψη ήταν ότι θα έπρεπε να έχουμε μια εύρωστη θέση, να πάμε στην Ολομέλεια, να έχουμε οντελή τη Ολομέλεια και κατόπιν να διαπραγματευτούμε. Και νομίζω ότι πάνω κάτω αυτό προτείνατε και εσείς κύριε Χερνέρ, αλλά τώρα όταν, κατά την επικοινωνία με τα άλλους θεσμούς, με τα άλλα οργανά, κατέστη σαφές σε μένα ότι θεωρούν τα άλλα οργανά ότι δεν είναι ευέλικτο το Κοινοβουλίο και δεν είναι έτοιμο να διαπραγματευτεί, αλλά αυτή δεν είναι η θέση μου. Ένα κράτος ε, μέλος που δεν είναι το δικό μου είπε ότι θα γίνει κηρύξη πολέμου αν πάμε στην Ολομέλεια με το φυστάμενο κείμενο. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την οδό. Έτσι λοιπόν προσπάθησα να εκπονήσω τροπολογίε που δείχνουν την εικονότητα του Κοινοβουλίου να συμβιβαστεί, να δημιουργηθεί κατάλληλη ατμόσφαιρα για τον τριμερή διάλογο και φυσικά η κανονική διαδικασία θα είναι να συναντηθούμε με όλε τι ομάδε ε, και με του συζητητέ στο Κοινοβούλιο και Φυσικά θα συζητήσουμε μεταξύ μα τι κόκκινε γραμμέ και θα πούμε στην τρομερή διάλογο κατόπιν να διαπραγματευτούμε τα υπόλοιπα όργανα. Και ακόμη με αυτέ τι τροπολογίε δεν προσποιούμε ότι είμαστε εδώ ε, στο παραπέντε μία συμφωνίας. Ε, Επίτροπος είπε ότι ε, μέχρι τα τέλη του Ιουνίου, που δυνάμει της ε, Προεδρία τη Δανία, θα μπορούσε να ολοκληρωθεί αυτό το θέμα, αν δείξει και βούλη στο Κοινοβούλιο, αν ε, δώσουμε το φακέλο στην Κυπριακή Προεδρία. Ε, δεν νομίζω ότι θα υπήρχαν ε, πολιτικές αντιρρήσεις, αλλά θα έπρεπε να ξαναρχίσουμε από την αρχή, να ξαναβρούμε το νήμα, ενώ οι Δανείοι είναι πάρα πολύ καλά ενημερωμένοι και έχουν μιλήσει με τα άλλα μέλη του Συμβουλίου. Κοιτάξτε, νομίζω ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια δυνατότητα να συμφωνήσουμε μέχρι τα τέλη Ιουνίου, αν το περάσουμε από την Ολομέλεια και έχουμε μια εντολή για να μπούμε σε διάλογο με τα υπόλοιπα όργανα. I would have a question to, to, to David Martin. Έχω μια ερώτηση για τον κύριο Μάρτιν. Ε, σπάνια μιλάτε και καταλαβαίνω τα όσα λέτε, αλλά δεν είμαι πεισμένος γιατί ε, συνήθως σας παρακολουθώ να σας πω γιατί δεν είμαι πεπισμένος. Πέρα πέραν του ίδιου του στόχου, όλοι συμφωνούμε ότι θα ήταν καλό να το προωθήσουμε το θέμα αυτό, να σημειώσουμε πρόοδο, αν είναι δυνατόν, ε, υπό την Προεδρία της Δανίας. Υπάρχουν ε, πολύ καλοί λόγοι να προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Όμω, ε, η ερώτησή μου είναι να μην χάνουμε χρόνο. Αν ε, τώρα πάμε στην Ολομέλεια και μόνο μετά την Ολομέλεια θα έχουμε εντολή για διαπραγμάτευση, θα έχουμε τη διαπραγματευτική ομάδα. Δηλαδή η Προεδρία της Δανίας εξαναγκάζει το Κοινοβούλιο να πάει τώρα στην Ολομέλεια αν δείξουμε ε, αυτή την καλή θέληση λοιπόν στη συζήτηση τώρα στην Επιτροπή και κατόπιν συστήσουμε μια ομάδα διαπραγματευτική και αρχίσουμε τις διαδικασίες στον τριμερή διάλογο. Μήπως ε, θα κινηθούμε έτσι πιο γρήγορα και θα πετύχουμε περισσότερα. Γιατί εγώ αυτά πιστεύω. Εσείς δεν με πείσατε, μήπως ε, θα μπορούσατε να με πείσετε. Δεν νομίζω ότι να συμβίβαστε τα δύο αυτά και ευχαρίστως ε, θα άρχιζαν τη συζήτηση και με τα υπόλοιπα όργανα αλλά ω ένα βαθμό επιζητώ και την εντολή, γιατί δεν θέλω να μπω σε διαπραγματεύσει με τα υπόλοιπα όργανα και κατόπιν ε, να δω ε, ότι δεν ξέρουμε τι ήθελε το Κοινοβούλιο. Έτσι λοιπόν η ψήφο στην Ολομέλεια θα είναι ένα τεστ για το πόσο μακριά είναι έτοιμο να προχωρήσει και το Κοινοβούλιο. Αλλά ε, ευχαρίστως να συνεχίσω τις συνδετικές συζητήσεις που έχω ήδη με Κομισιόν και Συμβούλιο και ευχαρίστως ε, να το εξηγήσω, αλλά υπάρχει και πρόβλημα ε, χρονοδιαγράμματος για την επόμενη εβδομάδα δεν έχουμε εργασίες και αν μπορούσαμε να έχουμε μια συνάντηση με τα υπόλοιπα όργανα πριν την Ολομέλεια, ευχαριστώ να προσπαθήσω να το οργανώσω. Ναι. Πολύ ευχαριστώ να συζητήσω με όποιον συνάδελφο, ό,τι ώρα, μέρα νύχτα, λίγο πολύ. Αλλά θα πρέπει και να γίνει συζήτηση και η ψηφοφορία. Εμείς ως Επιτροπή Συνταγματικών Θεμάτων έχουμε μια υποχρέωση που ίσως δεν βαρύνει άλλες επιτροπές, ότι πρέπει να είμαστε απόλυτα ε, διεξοδική και αυστηρή ως προς τις διαπραγματεύσεις. Και τουλάχιστον για τη δική μου ομάδα, μπορώ να σας πω, νομίζω ότι ισχύει για όλες τις ομάδες, ότι δεν θα παίρναγε πολύ εύκολα το να δώσουμε μια εν λευκό επιταγή στην Επιτροπή να προχωρήσει ε, στην κοινοβουλευτική μας επιτροπή να προχωρήσει χωρίς περιορισμούς για τη διαπραγμάτευση αυτή. Επομένω. Εάν θέλετε να προχωρήσουμε πριν από τις 2 Μαΐου, πολύ καλά, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει συζήτηση στην Ολομέλεια. Και με καλή προετοιμασία σε επίπεδο κοινοβουλευτικών ομάδων. Πρόεδρος. Λοιπόν, εγώ λοιπόν ε, θα δώσω μια ένδειξη αν ε, τον ε, Μάιο μπορέσουμε να συζητήσουμε στην Ολομέλεια το θέμα αυτό. Η Επιτροπή μας κατόπιν συνεδριάζει τις επόμενες ημέρες και μπορούμε να διορίσουμε την ομάδα που θα κάνει τις διαπραγματεύσεις στον τριμερή διάλογο. Δεν υπάρχει ε, ουσιαστικά κάποιο αμφίσιμο θέμα εδώ, κύριε Μάρτιν. Μπορούμε να το δρομολογήσουμε για το Μάιο. Αυτή είναι η πρόταση του εισηγητή. Νομίζω ότι δεν έρχεται σε αντίθεση με όσα είπε ο κύριο Έφνερ και νομίζω ότι και οι υπόλοιποι συμφωνούν και μπορούμε να περάσουμε στο θέμα που αφορά το πρωτόκολλο ε, για την τσεχική δημοκρατία. Έχουμε ε, εδώ ε, ουσιαστικά το θέμα της μη συμμετοχής στη σύμβαση. Ο κύριος Ντάφη είναι ο συγητής, το έχουμε ήδη συζητήσει αυτό. Αλλά δεν εγκρίθηκε η έκθεση Ντάφ. και στην τελευταία συνεδρίαση ακούσαμε τρεις βουλευτές από την Δημοκρατία. Και στο σημείο αυτό θα δώσω το λόγο στον κύριο Νταφ για να δούμε τι μπορεί να μας προτείνει για το πώς θα προχωρήσουμε στο θέμα αυτό. Που εμείς όμως το έχουμε um, Ευχαριστώ. Όπως ξέρετε, είχαμε πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων με τέσσερις Τσέχους συναδέλφους στο Στρασβούργο. Τους ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Που ήρθαν δηλαδή και ήταν έτοιμοι να συζητήσουν αυτό το θέμα μαζί μας και να εκθέσουν και την ε, διαφωνία που υπάρχει μεταξύ των πολιτικών κομμάτων στο Τσεχικό Κοινοβούλιο από αυτού. Πέρα από οτιδήποτε άλλο, με έπεισε για το ότι η δικιά μου προσέγγιση ήταν ορθή. Και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να εκφράσει αρνητική θέση όσον αφορά τη συμπερίληψη του πρωτοκόλου στη Λισαβόνα γιατί θα οδηγούσε σε νομική αβεβαιότητα και σε σύγχυση. Ίσως, μάλιστα, όπως εξήγησα και εξηγώ στην αιτιολογική έκθεση, ίσως δημιουργηθούν προϋποθέσεις όπου ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων τίθεται εν κινδύνο. Νομίζω ότι είναι καθήκον πρωταρχικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προστατεύσει και να προωθήσει την ακυρεότητα του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων και να ερμηνεύεται ομοιόμορφα στα δικαστήρια των χωρών μελών. Δεν πιστεύω, πως γνωρίζετε, ότι εφόσον οι Τσέχοι συμπεριληφθούν στο πρωτόκολλο Πολωνίας και Ηνωμένου Βασιλείου, δεν πιστεύω ότι θα γίνει τίποτα άλλο πέρα από το ότι θα τονιστεί η και οι κίνδυνοι που ελοχεύουν. Στη δεύτερη έκθεση έχω επεκταθεί ε, ουσιαστικά. Έχω διάφορες αιτιολογικές σκέψεις και μιλάω εκεί πιο άμεσα από ότι στην πρώτη μου έκθεση για τους λόγους για τους οποίους πιστεύω ότι πρέπει να καταλήξουμε στο συμπέρασμα αυτό. Ελπίζω οι συνάδελφοι να συμφωνήσουν για το ότι η επιχειρηματολογία μου ε, βασίζεται στα στοιχεία τα οποία έχουμε και στην ανταλλαγή απόψεων που είχαμε στο Στρασβούργο. Ο κύριος Μπροκ στην τελευταία συνεδρίαση πρότεινε αναβολή να μην προχωρήσουμε περισσότερο με την έκθεση αυτή. Να αφήσουμε την Τσεχία να προχωρήσει στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις και να τις παρακολουθήσουμε απλώς. Όμως δεν θα ήθελα να στηρίξω την ιδέα αυτή του Μπροκ. πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο μας οφείλει να γνωμοδοτήσει βάσει των συνθήκων. Και ότι ακόμα και αν μας πάρει χρόνο η γνωμοδότηση, πρέπει και πρέπει να είμαστε και πολύ προσεκτικοί στην προσέγγισή μας. να προχωρήσουμε χωρίς άλλη καθυστέρηση. Συνεπώς θα ήθελα να οριστεί προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών στη δεύτερη αυτή έκθεση. Και μετά να πάμε στην Ολομέλεια με την τακτική διαδικασία. Η σύσταση για συνέλευση ή όχι είναι ίδια. Όπως και την πρώτη φορά. Το μόνο που πρέπει να κοιτάξουν οι συνάδελφοι είναι το ψήφισμα. Ευχαριστούμε τον κύριο Ντάφ. Κύριε Προσμάτη. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνάδελφο κύριο Νταφ για την εξαίρετη αυτή έκθεση που παρουσιάζει νέες ιδέες και νέες προσεγγίσεις στην ε, ενημέρωση που λάβαμε την προηγούμενη φορά. Στα τελευταία μου ομιλία, στις παρουσιάσεις μου είχα μιλήσει για τον λεγόμενο αποκλεισμό ε, ε, εξαίρεση της ε, τσεχία. Ε, θα ήθελα να αναφερθώ τώρα στο πρωτόκολλο και φαίνεται ότι υπάρχουν αντικρουόμενες ε, νομικές πραγματογνωμοσύνες. Φαίνεται ότι η μία λέει ότι δεν υπάρχει καμιά επίπτωση ως προς την ανομετάξη της τσεχικής δημοκρατίας και η άλλη λέει ότι παρεμβαίνει το λόγο λόγω πρωτόκολλο στην ιστορική ένωμη τάξη και συμφωνώ με τον εισηγητή μα ότι μπορεί να προκύψει ασάφεια ω προ το τι ισχύει στο δικαίωμα. Χρειάζεται όμω για τον πολίτη ασφάλεια δικαίου και πρέπει να εξασφαλιστεί η προστασία των δικαιωμάτων του. Απεστάλλει από τα εμπορικά επιμελητήρια της Τσεχίας μια επιστολή στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού που επισημανόταν ότι έχει το ίδιο δικαίωμα κάθε άλλο πολίτη και ο Τσέχος πολίτης σε ασφάλεια δικαίου. Συμφωνώ λοιπόν με τον εισηγητή και ήθελα να πω και δύο λόγια για την ε, κατάσταση την πολιτική κατάσταση, γιατί διανύει την δέκατη πολιτική της κρίσης η κυβέρνηση. Αύριο πρόκειται να, δοθεί, να γίνει μάλλον ψηφοφορία για ψήφο εμπιστοσύνης. Το τρίτο μικρότερο κόμμα του συνασπισμού έχει αποτομηθεί σε δύο μικρότερες φράξεις, δηλαδή πολιτικές ομάδες. Ωστόσο βλέπουμε ότι η πλειονότητα αυτών, από ό,τι λένε οι εθνικοί βουλευτές, η πλειοψηφία μάλλον για την κυβέρνηση θα διατηρηθεί. Αλλά η κατάσταση είναι πάρα πολύ ρευστή, μέρα με τη μέρα αλλάζει και πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργό Νέτσα μπορεί ακόμη να χαίρει τη εμπιστοσύνη 102 έως 103 βουλευτών από τους άρα θα καλύψει τις 100 ψήφους που χρειάζεται για να διατηρηθεί στην εξουσία η κυβέρνησή του. Ευχαριστώ. Κύριο Σένιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η έκθεση αυτή αφορά μια πρόταση για το πρωτόκολλο που έχει προσαρτηθεί η Συνθήκη της Λισαβόνας για την τσεχική δημοκρατία σε σχέση με το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων που θέλουν οι Τσέχοι να ε, ενσωματωθεί πέραν μια διακήρυξη στην οποία έχουν προβεί. Ε, ο κύριος Ντάφ όμω λέει ότι δεν πρέπει να εξεταστεί αυτή η πρόταση. Εδώ έχουμε δύο ζητήματα όμω. Αν αρνηθούμε να εξετάσουμε αυτή την πρόταση τροποποίηση συνθήκε, θα ε, ισοδυναμούσε αυτό με μια απαράδεκτη απόρριψη τη εθνική ανεξαρτησία και εθνική κυριαρχία ενό κράτους μέλους. Και δεύτερον, θα αποδεικνύονταν για άλλη μια φορά η υποκρισία και η προσωπία τη Ευρωπαϊκή Ένωση που μα είχε άλλωστε αποδείξει ο Τόνι Μπλερ, γιατί μα είχε ξεκάθαρα πει ότι ότι έχουμε την δυνατότητα και παραθέτω τη ε, παρέκκληση για τα θέματα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών. Έτσι λοιπόν με την πρόταση αυτή για απορρίψη δυνάμει του, ε, του πρωτοκόλλου αυτού θα σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να εξαιρεθεί από την ισχύ του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων που άλλωστε έχει δοθεί Ω ερμηνεία από διάφορα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δηλαδή στο οποίο καταλήγει ο, Βρετανό, Βρετανός αλλά και κάθε άλλος πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι οι Βρυξέλλε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν είναι αξιόπιστα. Δεν πρέπει ποτέ να τα πιστεύουμε. Ευχαριστώ πολύ. Σεφλίν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και ευχαριστώ όλους όσοι έλαβαν μέρος στη συζήτηση αυτή μέχρι τώρα. Τίνω να συμφωνήσω με τα όσα είπε ο κύριο Νταφ για την αβεβαιότητα, για τη σύγχυση που μπορεί να επικρατήσει. Και δεν ε, θυμάμαι σε προηγούμενη περίσταση, στα χρόνια που έχω δώσει στο Κοινοβούλιο, να είχαμε αντιμετωπίσει τόσο πολλά προβλήματα και κίνδυνο σύγχυση και περιπλοκών. Υπάρχει λοιπόν αυτή η υποτιθέμενη παρέκκληση που δεν είναι, παρα, παρα, δεν είναι συγκεκριμένη παρέκκληση, αλλά δεν είναι και σίγουρο τι ακριβώ είναι. Το θέατρο του παραλόγου εν ολίγης. Και όπως έχω πει και άλλες φορές ε, πάνω στο ίδιο θέμα, τα πολιτικά και τα νομικά επιχειρήματα που θα μπορούσε κανείς να προβάλλει την προς διαφορετικές κατευθύνσεις και νομίζω ότι αυτό πρέπει να υπογραμμίσουμε και το πρόβλημα αυτό να το εξετάσουμε ε, ε, με το πρόκριμα ε, εάν επικρατεί η νομοθεσία έναντι της πολιτικής ή η πολιτική έναντι της νομοθεσίας, έναντι του δικαίου. Δεν έχω εγώ απάντηση να δώσω, και, αλλά πιστεύω ότι πράγματι αυτό είναι το επίκεντρο του ζητήματος. Εάν λοιπόν επικρατεί το δίκαιο έναντι της πολιτικής θα οδηγηθούμε σε περαιτέρω πολιτικά προβλήματα. Εάν όμως πούμε ότι επικρατεί πολιτική έναντι του δικαίου τότε προξενούμε ακόμη περισσότερη αβεβαιότητα, νομική και βέβαια σύγχυση. Γι' αυτό λοιπόν ε, μόνο προβληματισμούς αναφέρω, όχι λύσεις ε, και σε όσα είπε η κυρία Χάτα, νομίζω ότι ναι, όντω βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση η κυβέρνηση τη Τσεχία αυτή τη στιγμή. Ίσως όμως να είναι και η στιγμή να αποφασίσει, να κρίνει εάν προτιμεί μία πολιτική βεβαιότητα μέσα στη τσεχική δημοκρατία αυτή τη στιγμή και μπορεί η τωρινή κυβέρνηση να διατηρήσει την ε, πλειοψηφία της, ο τωρινός συνασπισμός, από την άλλη, ο Πρωθυπουργό Νέτσεστε έχει, δείξει, έχει δώσει αφή μηνύματα ότι δεν θέλει να συνεχίσει με συνασπισμό τριών, με, μάλλον με πλειοψηφία μόνο τριών ψήφων. Και ε, είναι ξεκάθαρο ότι αυτό προξενεί πολλά προβλήματα, δυσκολίε και επανέρχομαι στη λέξη ασάφεια και σύγχυση. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε κύριε Στασκόφσκι. Στο παρελθόν έχω τοποθετηθεί για το θέμα αυτό. Θα ξεκινήσω, Άντριο, όταν μεταξύ όταν μιλάμε για αυτά τα πρωτόκολλα. Εμένα δεν μου αρέσουν αυτά τα πρωτόκολλα, ούτε μου αρέσει η Πολωνία να είναι μία από τις χώρες που ζήτησε τέτοιο πρωτόκολλο. Και αν έδινα κάποια συμβουλή στην κυβέρνησή μου, θα τη συμβόλευα να ε, βγει εκτός του πρωτοκόλλου αυτού. Αυτή είναι η άποψή μου για το ίδιο το πρωτόκολλο. Παρ' όλα αυτά, όταν λέμε και ξέρουμε ότι αυτό είναι πολιτικό θέατρο, δεν έχει καμία σχέση με την διακύβευση του χάρτη, της χάρτας. Και αν κάποιος λέει, όπως είπε η συνάδελφος, ότι υπάρχουν αποκλίνουσε απόψεις, εγώ ουσιαστικά ακολουθώ όσο λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Και για μένα αυτό αρκεί. Λέει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα με την ομοιόμορφη εφαρμογή. Έτσι λοιπόν πιστεύω το δικαστήριο. Κάποιες φορές ε, μου αρέσει το όραμα του Άντριου για τις ξεκαθαρές λύσεις, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε τις ξεκαθαρές λύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι τόσο λεπτό αυτό το θέμα, δηλαδή ό,τι και να το ε, ε, θέμα της, των αρμοδιοτήτων, το θέμα Ε, του διαλόγου μεταξύ του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και του Συνταγματικού Δικαστηρίων. Ξέρετε λοιπόν ε, πόσο δύσκολο είναι αυτό το θέμα και γι' αυτό υπάρχουν ε, τέτοιες λύσεις, γιατί πολλές φορές είναι ξεκάθαρο να βρούμε σαφείς ξεκάθαρες λύσεις για τα πολιτικά αυτά προβλήματα. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πολιτικό θέατρο αυτό και αποδείχτηκε αυτό από τη συνάντησή μας με τους ε, τσέχου συναδέλφου Είναι πολιτική η συζήτηση αυτή, έχει συνταγματική και δεν θα πρέπει να συμμετάσχουμε σε αυτή γιατί θα δημιουργήσει μόνο προβλήματα για αυτό το κοινοβούλιο και μάλιστα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Έχουμε το δημοσιονομικό σύμφωνο που πρέπει να ακυρωθεί από τα κράτη-μέλη κτλ. Και ακόμη και αν ε, δεν συμφωνώ με τα κίνητρα, ε, για τα οποία, βάσει των οποίων ζητούνται αυτό το πρωτόκολλο μπορεί να δημιουργήσει μια λάθος ετύπωση ότι διακυβεύεται η χάρτα και τη ομοιόμορφη εφαρμογή. Και νομίζω ότι δεν θα πρέπει εμείς ε, ε, να θεωρηθεί ότι μπερδευόμαστε σε συνταγματικές ε, συγκρούσεις και είναι αυτό το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε αυτό. Και θα πρέπει να περιμένουμε να λυθεί αυτό από τους Τσέχους. Νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη λύση. Και να σας πω ότι συχνά δεν συμφωνώ με τον κύριο Άγνιου, αλλά όταν λέει ότι ακόμη και αν είναι λάθος, αλλά αυτή η ιδέα ότι υπόσχεται κάτι το Συμβούλιο σε ορισμένα κράτη-μέλη και στη συνέχεια υπαναχωρεί. Κοιτάξτε, θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη αυτό το επιχείρημα, να μιλάμε για το πλαίσιο και αν δείτε και τη συγκυρία είναι πραγματικά δύσκολη. Επαναλαμβάνομαι, το ξέρω, δεν είναι ότι μου αρέσει το πρωτόκολλο, δεν μου αρέσει. Και όπως είπα, δεν θα θέλω ούτως ή άλλως να υφίσταται τη δημιουργία σύγχυση. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν θέτει σε κίνδυνο τη χάρτα και αυτό είναι αμφισβήτητο. Αλλά το θέμα είναι τι θα κάνουμε εμείς. Αν εμείς ε, γινόμαστε κριτές ε, εσωτερικών ε, συνταγματικών συγκρούσεων. δεν θα ήθελα να αποτυπωθεί μια τέτοια εντύπωση γιατί νομίζω ότι είναι επικίνδυνο κάτι τέτοιο και μάλιστα γιατί και για το μέλλον θα υπάρχει πρόβλημα. Και τελικά αν είχα κάποια αμφιβολία ότι αυτό δεν θα επιλειόταν εσωτερικά, αν είχα αμφιβολία ότι θα έθετε σε κίνδυνο τη χάρτα. Θα διακύβευε τη χάρτα με οποιοδήποτε τρόπο. Ουσιαστικό θα σας υποστήριζα, αλλά δεν πιστεύω κάτι τέτοιο. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει ανάγκη εμείς να κάνουμε ένα τόσο δραστικό βήμα που θα μπορούσε να βλάψει την αξιοπιστία μας και θα μπορούσε ε, να καταστήσει την κύρωση του Δημοσιονομικού Συμφώνου ακόμη πιο επικίνδυνη από όσο είναι. Σας ευχαριστούμε. Μπρόντς. Ευχαριστώ. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην ε, περίπτωση του Αφγανού πολίτη ήταν το πρωτόκολλο 30, δεν αποτελούσε ένα opt-out η εξαίρεση, αλλά δεν είπε και τι ήταν είπε ότι δεν ήταν. Ορισμένοι πυρογνώμονε πρότειναν ε, ότι το νόημά του μπορεί να εξαρτάται από το αν ε, αφορά κάποιες συνθήκες ε, όπου αφαιρμόζεται μόνο η εθνική νομοθεσία ή πιθανόν όπου η νομοθεσία όπου μάλλον η Εθνική Νομοθεσία εφαρμόζει το κοινοτικό δίκαιο. Μπορεί να εξαρτάται από τις περιπτώσεις δηλαδή. Τώρα η εθνικη νομοθεσια εφαρμοζει το κοινοτικο δικαιο μπορει να εξαρταται τις περιπτωσεις δηλαδη τωρα η συναντηση με τους τσέχους βουλευτές ήταν ενδιαφέρουσα αλλά βέβαια αφορούσε περισσότερο την εσωτερική διαμάχη στη Τσεχική Δημοκρατία για το αν είχε δίκιο ή όχι ο πρόεδρος της Τσεχίας να ζητήσει το πρωτόκολλο 30 και όχι ε, επί των γεγονότων επί της ουσίας. Έτσι λοιπόν εμείς ήμασταν θεατές. Τώρα, ε, το, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, η κυβέρνηση της Πολωνίας και ο πρόεδρο της ε, Τσεχίας και η κυβέρνηση της Τσεχίας ε, ε, πίστευαν ότι οδηγήθηκαν να πιστεύουν ότι είχαν κάποιο είδους εξαίρεση ένα opt-out και άλλα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τότε που δεν είχαν μια διακριτή ταυτότητα τότε, ε, ήξεραν ότι το πίστευαν αυτό ή προσποιούνταν ότι το πίστευαν και επέτρεψαν ε, να παγιωθεί αυτή η πεποίθηση. Έτσι λοιπόν ε, το ερώτημα παραμένει. Ποιος είναι η πηγή, ποιος είπε ε, ότι ε, είσαι κάτι τέτοιο. Ένας τρόπος ε, να βγούμε από αυτό είναι να έχουμε ένα πρωτόκολλο. Βέβαια, ε, έχουμε και το δεύτερο ερώτημα που έρχεται. Ποιος ουσιαστικά συνέταξε το πρωτόκολλο αυτό και ποιε συμβουλές δόθηκαν για τη σύνταξη αυτού του πρωτοκόλλου. Επίσης πρέπει να θυμόμαστε ότι δόθηκε μία διαβεβαίωση στο Κοινοβούλιο του Ευρωπαϊκού του Ηνωμένου Βασιλείου όταν ε, κυρώθηκε η συνθήκη της Λισαβόνας. Ε, η κύρωση ε, όταν υλοποιείται το Κοινοβούλιο επετεύχθη από μία μη αλήθεια. Δεν μιλώ για ψέμα, δεν ξέρουμε αν ο τον Ιμπνερή ήξερε ότι ήταν αλήθεια, πίστευε ότι ήταν αλήθεια, υποψίαζε ότι μπορεί να μην ήταν αλήθεια, αλλά φαίνεται ότι ήταν κάτι μη αληθές. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν έχει την ικανότητα να δίνει ε, κάποιες διαβεβαιώσεις για τις συνθήκες τις οποίες συμφωνεί και πάλι έρχεται εδώ το θέμα στις διαπραγματεύσεις με την Κροατία. Δόθηκαν διαβεβαιώσεις από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην Κροατία και όλα αυτά εγγραφόταν στο πρωτόκολλο. Δεν μπορώ να απαντήσω αυτήν την ερώτηση. Τώρα σε ό,τι αφορά Μακεδονία, Σερβία και άλλες χώρες... Ε, που έχουν ζητήσει την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δίνονται και σε αυτές κάποιες εγγύσεις και αυτές ε, οι εγγύσεις, οι διαβεβαιώσεις που δίνονται έχουν κάποια αξία. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπρακ είναι εδώ μαζί μας. Είναι παρατηρήτρια. Δεν πρόφερα καλά το όνομά σας, με συγχωρείτε. Είναι παρατηρήτρια για την Κροατία και είναι η πρώτη φορά ε, αυτή την ε, επιτροπή. Σας έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα... Θα μιλήσω αγγλικά και μπορώ να μιλήσω ιταλικά. Καταρχήν, σας ευχαριστώ για το πόσο καλά μας καλωσορίσατε, την άνθρωπο καλωσόρισμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε αυτή την Επιτροπή. Είμαι πάρα πολύ ε, ευτυχής που συνεργάζομαι μαζί σας. Δεύτερον, θέλω να ευχαριστήσω όλα τα κοινοβούλια των κρατών μελών που ήδη κύρωσαν ε, την συνθήκη προσχώρησης. Για την Κροατία έξι χώρες ήδη το έπραξαν ε, και τις ευχαριστούμε για την ταχεία διαδικασία και είμαστε πεπισμένοι ότι η διαδικασία αυτή θα κύλησε ομαλά μέχρι την 1η Ιουλίου του χρόνου όταν θα προσχωρήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα πρωτόκολλα για τη Τσεχία συνδέονται κατά κάποιο τρόπο Πώς λέγεται το έγγραφο. Ψήφισμα. Λοιπόν, αναφέρομαι στο σημείο, δηλαδή αυτό συνδέεται με τη συνθήκη προσχώρηση τη κροτίας, αλλά χθε η Γερουσία στη Τσεχία κύρωσε την συνθήκη προσχώρησή μα, αλλά δεν νομίζω ότι έχουμε πλέον αυτό το πρόβλημα. Χθε ομόφωνα η Γερουσία στη Τσεχία κύρωσε τη συνθήκη προσχώρηση της Κροατία. 259 βουλευτέ ήταν παρόντες και όλοι συμμετείχαν στην ψηφοφορία ε, υπόθηκε ότι το κάτω τμήμα του Κοινοβουλίου Κατουβουλή Βουλή πρόκειται, της Τσεχίας πρόκειται πολύ σύντομα να επικυρώσει την συνθήκη προσχώρησης της Κροατίας για την παρακολούθηση. Η έκθεση παρακολούθησης ε, δημοσιεύτηκε προ, λίγο ημερών από την Κομισιόν και ήταν αρκετά θετική αν μπορώ να τοποθετηθώ, αλλά δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα το κρίνουμε αυτό. Τον Οκτώβριο αναμένουμε την πλήρη έκθεση παρακολούθησης και Πιστεύουμε και ότι και αυτή θα είναι θετική. Γνωρίζουμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε με τις μεταρρυθμίσεις μας, καθώς είμαστε η πρώτη χώρα που έκανε τις διαπραγματεύσεις ανά κεφάλαια και ανά ε, κριτήρια σύγκρισης. Κράτησαν πολλοί διαπραγματεύσεις, όμως είμαι βέβαιη ότι θα είναι θετική η έκθεση του Οκτωβρίου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Έφνερ. Σε αυτή τη δύσκολη συζήτηση. Με χαρά ακούμε ότι υπάρχουν και κράτη-μέλη στα οποία βαίνουν χωρίς δυσκολίες τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν για τόσο μας την Κροατία. Θα ήθελα πάντως εγώ να πω ότι αισθάνομαι σχέση με το πρωτοκόλλο αυτό όλο και πιο αμήχανα γιατί έχουμε βρεθεί ως Κοινοβούλιο και ως Επιτροπή σε μια όντως πολύ περίπλοκη κατάσταση, άθελά μας, μας οδήγησαν στην κατάσταση αυτή. Και πάντα βέβαια πρέπει να είναι οι κανόνες και διατάξεις αφής, αξιόπιστοι, να είναι κάτι πάνω στο οποίο κανείς να μπορεί να οικοδομήσει και όχι ε, καλά μια στον κάπο και να γίνουν από μια μεριά και από την άλλη. Τώρα λοιπόν ε, καλό θα ήταν να ξεκαθαρίσει το τι τελικά θα ισχύει στη Τσεχία και αυτό που θα ισχύσει να αντιστοιχεί και στη βούληση του τσεχικού λαού. Οι δύο ε, βουλές της ε, Τσεχίας κύρωσαν την συνθήκη της Λισαβόνας χωρίς επιφύλαξη, δείχνοντας αυτή την εμπιστοσύνη. Ο πρόεδρος διατύπωσε επιφύλαξη, που δεν είχε συζητηθεί και συμφωνηθεί από τα κοινοβούλια. Το θέμα είναι ποιον πρέπει να ακολουθήσουμε τώρα. Ένα δίδαγμα το οποίο μπορούμε να αποκομίσουμε είναι ότι δεν μπορεί κανείς τόσο έλαφρα την καρδία να επιτρέπει ε, την εισαγωγή επιλογών opt-out ή opt-in, ε, αποκλεισμού από συνθήκες και από συμβάσεις. Νομίζω ότι παρά ήταν ε, γρήγορη η δυνατότητα που δόθηκε στην ψυχία για αποκλεισμό, χωρίς συζήτηση, χωρίς ε, διατύπωση των συνεπειών. Και τώρα η μεγάλη δυσκολία είναι το τι θα πράξουμε. Το Κοινοβούλιο πιστεύω ότι οφείλει και πρέπει να τοποθετηθεί. Θα μπορούσαμε να πούμε βεβαίως ότι απέχουμε. Δεν εμπλεκόμαστε στην υπόθεση αυτή, αλλά ισοδυναμούσε με ε, μη τήρηση των δεσμεύσεων και των υποχρεώσεων που έχουμε στην υπόθεση αυτή. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει να τοποθετηθούμε. Και να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι δεν βλέπουμε κανένα λόγο για κύρωση του πρωτοκόλλου αυτού. Όλα τα άλλα ξέρω ότι τα έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν, δεν θα τα επαναλάβω λοιπόν ως προς, προς την ουσία. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Γκολτιέρη. Ευχαριστώ. Είμαι σύντομος. Μια παρατήρηση μόνο θέλω να κάνω για το θέμα της δέσμευσης του Συμβουλίου και το ρόλο του Κοινοβουλίου. Το Κοινοβούλιο έχει ένα ρόλο συμβουλευτικό και αυτό δεν είναι τυχαίο. Έτσι λοιπόν, ο συμβουλευτικό χαρακτήρα ε, τη γνωμοδοτησή μα μα απελευθερώνει και πολιτικά από δεσμεύσει. μπορούσαμε βέβαια να έχουμε και ένα πιο ισχυρό ρόλο, αλλά είναι σαφέ ότι ακριβώ επειδή ο ρόλο μα είναι συμβουλευτικό, δεν είναι δεσμευτικό. Έτσι λοιπόν το Συμβούλιο, οι κυβερνήσει μπορούν να προβαίνουν σε δεσμεύσει γιατί είναι σε θέση να προχωρήσουν με τα δικά του εθνικά κοινοβούλια. Ακριβώ γιατί το κοινοβούλιο πρέπει να γνωμοδοτήσει. Δεν βλέπω εγώ να υπάρχει πρόβλημα λοιπόν. Έτσι λοιπόν εμεί μπορούμε ελεύθερα να εκφράσουμε την απόψή μας και όπως γνωρίζετε είναι αρνητική για τη δική μας ομάδα. Όπως είπε και ο συνάδελφος ε, Νταφ, είναι ε, σαφές ότι δεν μπορούμε να καθυστερούμε Επαόριστον πρέπει να την ε, υλοποιήσουμε αυτή τη γνωμοδότηση. Πρέπει να τοποθετηθούμε. Όμως, κατάλαβα καλά, οι συνάδελφοι του ΕΛΚ δεν ζητούν να μην δοθεί η γνώμη αυτή. Απλώς ε, ζήτησαν να έχουμε περισσότερο χρόνο για να σκεφτούμε το πράγμα και να δούμε και ποιες ε, είναι οι άμεσες εξελίξεις στην Τσεχική Δημοκρατία. Εγώ προσωπικά νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε. Κρίνω θετικά και το νέο κείμενο που μας πρότεινε ο συνάδελφος. Νομίζω ότι όταν ε, ορίσουμε το χρονοδιάγραμμα θα μπορούσαμε να λάβουμε θετικά υπόψη και την απέτηση να μην προχωρήσουμε με υπερβολική ταχύτητα. Δηλαδή μέσα στα όρια, τα κανονικά που έχουμε για περιθώριο λιγμών, θεωρώ ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη θέση που εκφράζεται από το ΕΛΚ. Μάλιστα. Ο κύριος Νταφ. Ευχαριστώ πολύ. Και ιδιαίτερα στην κυρία Φρουμπάτ. Για την παρθενική τη ομιλία εδώ. Ιδιαίτερα μας εντυπωσιάζει η πρόοδος που σημειώνει η Κροατία. και σε κανένα σημείο τη διαδικασία εδώ στην Κοινοβουλευτική μα Επιτροπή δεν συνδέουμε την ε, συνθήκη τη της Κροατία με το πρωτόκολλο για την Τσεχία. Ξέρετε ότι το πρόβλημα ήταν στο επίπεδο του Συμβουλίου. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να αντιδράσουμε μόνο. Για τον κύριο Μπρόνς. Η διατύπωση του πρωτοκόλλου για την αρμοδιότητα της διακυβερνητικής διάσκεψης, όχι του Συμβουλίου. αλλά της διάσκεψης, της διακυβερνητικής διάσκεψης, οποία επεξεργάστηκε την συνθήκη της Λισαβόνας. Τον κύριο Μπλερ δεν τον εκπροσωπώ, ούτε τον εκπροσώπησα ποτέ, ούτε καν τον ψήφισα ποτέ. Μάλιστα την εποχή, εκεί, την εποχή εκείνη είχα εκφράσει και είχα δημοσιεύσει σε άρθρο τις θέσεις μου για το πρωτόκολλο αυτό σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν απέκρυψα τις θέσεις μου. Αντιλαμβάνομαι ότι ορισμένοι τα πράγματα βλέπουν πιο πολύ άσπρο ή μαύρο. Εγώ βλέπω διάφορες διαβαθμίσεις του γκρίζου απόχρωση αχλής. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι έχουμε καθήκον ως Κοινοβούλιο να εποπιστούμε τις ευθύνες που έχει προσδιορίσει η συνθήκη και να βοηθήσουμε τους Τσέχους να καταλήξουν σε μια απόφαση, σε μια θέση για την υπόθεση αυτή. γιατί καταρχήν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να τοποθετηθεί για το αν θα εγγραφεί αυτό το πρωτόκολλο συνθήκη Τσεχία και μετά τα 27-28 τώρα κράτη-μέλη με τα εθνικά του κοινοβούλια. Άρα, ας μην ε, ε, υπερβάλλουμε τη σημασία που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην υπόθεση αυτή, αλλά ας μην την υποβιβάζουμε κιόλας. για το Ραφαέλ. Εγώ δεν είμαι δικαστήριο ούτε και δήλωσα ποτέ ότι δεν υπάρχουν δυσκολίε ως προς την ομοιόμορφη εφαρμογή του χάρτη. του Λονδίων, όπως είπε ο κύριος ε, Μπρόνς, ε, το δικαστήριο έχει επιφυλάξει πολλές φορές διατυπώσει ω προς την εφαρμογή του πρωτοκόλου και στην δεύτερη έκθεση. Προτείνω να πούμε ότι εάν το πρωτόκολλο ερμηνευθεί Ω προ το πεδίο και τι διατάξει του χάρτη, ότι ισχύει ω προ το πεδίο και τις διατάξει του χάρτη, θα έχει συνέπειε αρνητικές. Δεν είναι δεδομένο ότι θα ερμηνευτεί έτσι όμω. Υπάρχει κίνδυνο ωστόσο και θα πρέπει να τον αναγνωρίσουμε. Εγώ θα πρότεινα να, να ορίσουμε μια προθεσμία κάπου το καλοκαίρι, τον Ιούνιο ίσως, μια κατάθεση τροπολογιών, η οποία θα έχει σε συνέπεια η συζήτηση στην Ολομέλεια να εξαχθεί κάπου το φθινόπωρο. Και έτσι μέχρι τότε θα έχει πιστεύω ε, ξεκαθαρίσει και η πολιτική κατάσταση στην Τσεχία και θα έχουμε και εμείς περισσότερο περιθώριο να κατασταλάξουμε. Γι' αυτό, Πρόεδρε, προτείνω προθεσμία για τις τροπολογίες να οριστεί τον Ιούνιο. Eh, λοιπόν, ουσιαστικά μου πρότεινα η Γραμματεία ημερομηνία για τις τροπολογίες 10 Μαΐου για να ψηφίσουμε στη συνέχεια στις 30 Μαΐου. Εσείς προτείνετε μεγαλύτερη προθεσμία. Θα έπρεπε να είναι στις 24 Μαΐου για την παρουσίαση τροπολογιών και να ψηφίσουμε στις 19 Ιουνίου. Εκτός μικροφώνου το σχόλιο του κ. Γκουαλτιέρη. Νόμιζα ότι είπατε κάτι άλλο. Κύριε Ντάφε, εσεί τι θέλετε, θέλετε τη ψηφορία πότε. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Ε, ε, τον Ιούνιο είναι η προθεσμία. Οπότε θα έρθει το θέμα στην ε, Επιτροπή μας τον Ιούλιο και η Ολομέλεια θα ψηφίσει κάποια στιγμή το φθινόπωρο. Se gli altri colleghi sono d'accordo. Αν συμφωνούν οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Possiamo stabilire il termine per gli emendamenti. Μπορούμε να θέσουμε ω προθεσμία για τι τροπολογίε τη 14η Ιουνίου και κατόπιν θα ψηφίσουμε όταν είναι δυνατό. resta stabilito. Μάλιστα, το καθορίσουμε και αυτό. Έχουμε προχωρήσει αρκετά στην ημερησία διάταξη. Και τώρα έχουμε τον συνάδελφο Μέσσερ Σμιτ. Δεν είναι εδώ που θα μας μιλήσει σχετικά με τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θέλετε το λόγο, παρακαλώ. Thank you, Well, as you all know... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως γνωρίζετε όλοι, μου ζητήθηκε από την Επιτροπή μας να ετοιμάσω τη γνωμοδότηση αυτή για την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για την 28η ετήσια έκθεση, δηλαδή σχετικά με τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει ετοιμαστεί λοιπόν, είναι στο σημείο 17, θα βρείτε τη γνωμοδότησή μου. Θέλω όμως να σας αναφέρω μερικά κύρια σημεία της. Παράγραφος 2 Εδώ εκφράζουμε την λύπη μας για το ότι παρά τις μάτες προσπάθειες που κατέβαλαν Κοινοβούλιο και Επιτροπή να περιλάβουν τις οδηγίες δεσμευτικές διατάξεις, δεν τα καταφέραμε. Εγώ πιστεύω ότι οι δεσμευτικές διατάξεις έχουν άμεση σχέση με την τήρηση των προθεσμών και με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Γι' αυτό θα έπρεπε να συμπεριληφθεί κάτι τέτοιο ιδίω για την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Τα τεχνικά θέματα και οι λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με τις συνθήκες. Παράγραφος 4 τώρα. Εδώ επισημαίνω την σημασία που έχει η διαφάνεια στις δυστυχώς πάρα πολλές διαδικασίες επί παραβάση σε βάρος των χωρών ε, μελών, είτε επειδή δεν τρούν τις προθεσμίες, είτε δεν το κάνουν καλά, δεν ενσωματώνουν τις οδηγίες κλπ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τώρα πρέπει να παίξει ένα ρόλο κλειδί σε όλη αυτή τη διαδικασία. Πρέπει δηλαδή να ενημερώνεται κάθε φορά που υπάρχει μια τέτοια διαδικασία επί παραβάση για να μπορεί να αναλάβει το ρόλο του. Έπειτα στην παράγραφο 5 επειδή ακριβώ είναι πολύ σοβαρό το θέμα, εγώ και ελπίζω να συμφωνείτε, λέω ότι δεν πρέπει την παράβαση της μη ενσωμάτωσης μιας οδηγίας να την θεωρούμε ισοδύναμη με οποιαδήποτε άλλη παράβαση. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να φαίνεται γιατί καταλαβαίνετε ότι για το βιομηχανικό κλάδο ή για οτιδήποτε, μια χώρα η οποία δεν έχει ενσωματώσει μια οδηγία, καταλαβαίνετε ότι βάζει τις υπόλοιπες σε μειονεκτική θέση. Τέλος, στην παράγραφο 6 υπογραμμίζω ότι πρέπει να γίνεται ο σχετικός έλεγχος ομαλά, και σε περίπτωση ένα κράτος μέλος δεν έχει μπορέσει να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του, με τη ε, βάση των αποφάσεών μας, να μπορεί να υπάρχει δυνατότητα αγκαίρης παρέμβασης. Αυτές είναι οι προτάσεις μου και από εκεί και πέρα περιμένω τις δικές σας ιδέες, τροπολογίες και ελπίζω όλες οι πολιτικές ομάδες στο τέλος να στηρίξουν την γνωμοδότηση αυτή ό,τι παρατηρήσεις έχετε είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκολτιέρη. Πολύ σύντομα, εκ μέρου ε, τη ε, Σκιώδου, κυρίας τη κυρία Νέγκνερ, που δεν μπορούσε να παρευρεθεί σε αυτή τη συνεδρίαση. Να κάνω ένα θετικό σχόλιο για αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης η σκιώδης εισηγητρία επιφυλάσσεται βέβαια να ε, τοποθετηθεί περαιτέρω εις βάθος για την παράγραφο 8 σχετικά με τη δυνατότητα να έχουμε κανονισμούς αντιοδηγιών. Αλλά γενικά ε, κρίνει θετικά την γνωμοδότηση αυτή. Ευχαριστώ. Μάλιστα αν και ε, σκοτήσω του ΕΛΚ ε, δεν είναι εδώ, πρέπει να πάει στη Βραζιλία. Έτσι λοιπόν το λόγο έχει ο κύριος Νταφ. Ευχαριστώ. Θα το κοιτάξω από κοντά το θέμα και με κάθε σεβασμό όπως το αξίζει. Θα ήταν όμως νομίζω καλό αν είχαμε μπορέσει να συζητήσουμε αυτό το θέμα με τον Επίτροπο Σεύκοβιτς χτες. Μια ανταλλαγή απόψεων ήταν η χθεσινή που πιστεύω ότι δεν ήταν τόσο δυναμική ούτε και τόσο καρποφόρα για μας ή για εκείνον. Θα ήθελα λοιπόν η Επιτροπή να αντιδρούσε στην ε, πρόταση αυτή. Να μας πει τη γνώμη της δηλαδή, εν ευθέτω χρόνο. Σε μια άλλη συνεδρία, στην επόμενη συνεδρίασή μας προφανώς. Θέλετε να απαντήσετε παρακαλώ κύριε Μέσερσον. Ναι. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας. Στον κύριο Κολτιέρη θέλω να πω ότι γνωρίζω ότι μπορεί να είναι επίμαχη παράγραφος 8 ε, που μιλάει για περισσότερους κανονισμούς αντί για οδηγίες. Αλλά τι να κάνουμε, τα κράτη-μέλη από ό,τι φαίνεται δεν τα φέρνουν πέρας με τις οδηγίες. Και τα θεσμικά όργανα πρέπει να δράσουν κατάλληλα. Αλλά μπορούμε να το διατυπώσουμε κάπως διαφορετικά. Φυσικά χαίρομαι πάρα πολύ που η γενική αντιμετώπιση είναι θετική Μπορούμε να ξανασυζητήσουμε όλου του παραγράφου με του και ηγητέ, άμα θέλετε. Τώρα κύριε Ντάφ, συμφωνώ για αυτό που λέτε για τη συνάντηση με τον κύριο Σιεκόβιτ ε, Χτέ για το ότι πρέπει να έχουμε την άποψη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ναι, αλλά από την άλλη μεριά πρόκειται για γνωμοδότηση ε, πάνω σε μία έκθεση, η οποία γίνεται πάνω σε έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οπότε δεν ξέρω τι θα βγάλουμε αν ρωτούσαμε τον Σέκοβιτς. Για μένα ευχαρίστω να έχουμε συναντήσεις με τον Επίτροπο, αλλά ίσως θα ήταν καλύτερα εμείς οι σκιώδεις, όταν έχουμε καταλήξει σε μία θέση, τότε, ίσως πριν την ψηφοφορία, τότε να συναντηθούμε τον Σφέκοβιτς και να δούμε Μήπως ε, μπορεί τότε να μας βοηθήσει. Αυτό θα ήταν το καλύτερο νομίζω ο συμβασμό. Πάντως, στο στάδιο που βρισκόμαστε τώρα, που είναι αρχικό, είναι πιο σημαντικό να ακούσουμε τι λένε οι πολιτικέ ομάδε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπρόνς. Δεν θα μακρηγορήσω, αλλά δεν θα πρέπει και τη σιωπή μου να τη θεωρήσετε κατάφαση. Εντάξει, εγώ προτιμώ τι οδηγίες από του κανονισμού, γιατί οι κυβερνήσει μπορούν να παρακούσουν, μπορούν δηλαδή νομικά ε, τουλάχιστον ε, να το αντιμετωπίσουν διαφορετικά. Και όσο περισσότερο παρακούν, τόσο το καλύτερο. Ε, είσαστε πολύ συνεπεί με τον εαυτό σα, κύριε Μπρούντζα. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε τώρα. Νομίζω ότι αν θέλουμε να ψηφίσουμε στις 30 Μαΐου να παρουσιαστούν οι τροπολογίε μέχρι τις 10 Μαου. Ο κύριος Μέσσερ Σμιτ συμφωνεί. Μάλιστα. Δεν λένε υπάρχουν και άλλες αντιρρήσεις, συμφωνούν και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα το σημείο 18, τροποποίηση του άρθρου 123 του κανονισμού του Κοινοβουλίου σχετικά με τις γραπτές δηλώσεις. Ο κύριος Σταρκόφσκι είναι ο εισηγητής, συζητήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου λάβαμε 64 τροπολογίες και πριν να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία που προβλέπεται για τις 30 Μαΐου συμφωνήσαμε να ακούσουμε την άποψη του κυρίου Ταρκόφσκη για τις τροπολογίες και ενδεχομένως και το τι πιστεύουν και τα υπόλοιπα μέλη αυτής της Επιτροπής. Παρακαλώ κύριε Ταρκόφσκη. Κυρίε και κύριοι, καταρχάς σας ευχαριστώ θερμά για τις τροπολογίες σας. Η άποψή μου για τις γραπτές δηλώσεις παραμένει αρνητική. Ξέρετε και το έχω πει ξεκάθαρα ότι τον όρο καταργώ, καταργούνται, τον έχω συμπεριλάβει προκειμένου να προξενήσω συζήτηση, διάλογο. Δεν είναι αυτό το αποτέλεσμα στο οποίο το οποίο αποσκοπώ, στο οποίο αποσκοπώ τουλάχιστον όχι άμεσα. Αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να ε, συζητηθεί ιδιαίτερος και να εξορθολογιστεί ο ρόλος και η λειτουργία των κρατών δηλώσεων. Ίσως θα πρέπει να βρούμε μια διαφορετική διατύπωση στην επιχειρηματολογία μας. Έτσι λοιπόν όλες οι τροπολογίες οι οποίες στόχο έχουν να τροποποιήσουν πλήρως το μήνυμα της εκθέσεως και που προσπαθούν να ισχυριστούν ότι είναι πολύ ωραίε οι γραπτές δηλώσεις, είναι ένα εργαλείο που θα πρέπει διαρκώ να χρησιμοποιούμε, ότι δεν παρουσιάσουν καμία δυσκολία ή πρόβλημα και ότι απλώς η προβλημα και οτι απλω η επιτροπη δεν τι έχει τήρησει όπως θα έπρεπε, με βρίσκουν αντίθετο. Όπω είπα πρέπει να εξορθολογιστεί η χρήση του. Βεβαίω μπορούμε να συμφωνήσουμε, να συζητήσουμε συγκεκριμένε προτάσει. ε, παραδείγματι εκεί που λέμε ότι έχουν προσφέρει, αλλά δεν προσφέρουν πλέον επαρκώς, εγώ σημειώνω ότι έχουν μια κάποια αναξία ως εργαλείο που προξενεί, ε, που ανοίγει μια συζήτηση για ορισμένα θέματα. Μια συνετική λοιπόν προσέγγιση ως προς την αξιολόγηση του μέσου μπορεί να με βρει σύμφωνο, αλλά όχι πλήρης τροποποίηση του κειμένου. Διατηρούν λοιπόν μια κάποια αναξία, άλλωστε πρέπει να τις εξορθολογήσουμε. Και το πιο σημαντικό είναι να εξετάσουμε και πάλι τη διαδικασία, γιατί ξέρετε γίνεται ηλεκτρονικά, να δούμε πώς μπορούμε να τις προβάλλουμε, γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί πολλούς συναδέλφους. Η πρόταση του κ. Ταφ, που όμως είδαμε και σε άλλα σημεία, ότι θα πρέπει να δίνετε άδειο για την ε, πρόταση, για την αγαπητή δήλωση δηλαδή, μου φαίνεται ελκυστική. Αν και διαπιστώνω, Άντριου, μια αντίφαση στα όσα λες. Δηλαδή, αφενός με ένα, είσαι λιγότερο αρνητικό για, τι γραπτή, για τις δηλώσεις. Αφετέρου όμω μόλι ότι, δεν θα, πρέπει να δεσμεύουν το κοινοβούλιο. Αυτό δεν το αντιλαμβάνομαι. Εγώ είμαι υπέρ του περιορισμού του πεδίου του, του εξορθολογισμού. Εγώ προσπαθώ να δείξω ότι μπορούμε να έχουμε άλλα πιο χρήσιμα μέσα για να εξυπηρετήσουμε τον ίδιο στόχο. Αλλά εάν διατηρηθούν αυτέ οι γραπτέ δηλώσει και αν τι υπογράφουν πάνω από του μισού ε, βουλευτέ, τότε θα πρέπει να είναι δεσμευτικέ. Αλλιώ τι νόημα έχουν. Εάν λοιπόν μπορώ να πω, εντάξει, να καταλήψω τον όρο ε, καταργούνται, αν και ελπίζω ότι αυτό θα προξενήσει μια κάποια συζήτηση για το τι θα γίνει περαιτέρω. Αν εγκαταλείψω λοιπόν τον όρο καταργούνται και πω εντάξει διατηρούμε αλλά δεν είναι δεσμευτικές, τότε νομίζω ότι χάνει ακόμη περισσότερο νόημα όλο αυτό το εγχείρημα. Πρέπει να αποφασίσουμε αν είμαστε υπέρ του ενός, της μίας ή της άλλης λύσης και για τον εξορθολογισμό. Πολύ βεβαίω, ε, πολύ ευχαριστώ να κοιτάξουμε το θέμα τη ε, χορήγηση άδεια, δηλαδή να ενισχύσουμε το ρόλο του Προέδρου του Κοινοβουλίου ή να συζητήσουμε πόσοι θα πρέπει να είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να δώσουν υπογραφή σε μια γραπτή δήλωση, γιατί ακούγονται διάφορε προτάσει. μπορούμε να το συστήσουμε αυτό, αλλά μια πρόταση που ακούω από τον Ρομπέρτο Φερρυπίν ε, που παραπέμπει σε άλλα πιο σοβαρά μέσα, Φερρυπίν το δικαίωμα πρωτοβουλία, μου φαίνεται πιο αξιόπιστη. Και εδώ έρχομαι στο πιο αντιφατικό ζήτημα που θα πρέπει περαιτέρω να συζητήσουμε. Διότι ένας εύκολος τρόπος θα ήταν να πούμε σε μια μονοπαράγραφο ότι προσπαθούμε να ε, περιορίσουμε και να εξορθολογήσουμε τη γραπτή δήλωση, όχι γιατί θέλουμε να απεμπολίσουμε τη δυνατότητα για τα βουλευτές να κάνουν κάτι σε ένα θέμα σημαντικό και ένα θέμα το οποίο κατά τα άλλα όμως ε, οι πολιτικές ομάδες δεν υποστηρίζουν ή δεν είναι μεγάλης ε, απήχησης. Αλλά από την άλλη θέλουμε να υπογραμμίσουμε ότι υπάρχει το δικαίωμα πρωτοβουλία. Δηλαδή και προβάλλουμε αυτή τη δυνατότητα, λέμε γιατί τη διατηρούμε, γιατί υπάρχει, διότι χάρη στη συνθήκη έχουμε εξασφαλίσει περισσότερα μέσα και πάνω απ' όλα πιο ε, αποτελεσματικά μέσα για να δρούμε εκ μέρου των βουλευτών. Αυτή θα ήταν λοιπόν η light έκδοση, μία μόνο παράγραφο που δεν θα οδηγούσε, δεν θα απαιτούσε περισσότερε τροποποίησεις προς τον κανονισμό, ενώ μια πιο φιλόδοξη γραμμή θα ήταν ε, να ε, θεσπιστεί, να δημιουργηθεί ένα σύστημα και θέλω να το πω ε, έτσι ώστε να μην προσβάλλω κανέναν, ναι, μέσα από το οποίο μόνο οι σοβαρές εντό εισαγωγικών γραπτές δηλώσεις θα μπορούσαν να μεταγραφούν ως ε, πρωτοβουλίες ε, ως κείμενα του δικαίωματος πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου. Άρα μόνο εκεί όπου βλέπουμε ότι μια γραπτή δήλωση συνάδει με τη συνθήκη, με τα άρθρα της συνθήκης κλπ μπορεί να μετατραπεί σε δικαίωμα πρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου. Σε έκθεση πρωτοβουλίας. Ε, αυτό νομίζω είναι το πιο ελκυστικό και ενδιαφέρον στοιχείο που ακούγεται και ίσως θα πρέπει να μας απασχολεί στο πώς θα το υλοποιήσουμε. Άρα, εγώ θα ήθελα να ενισχυθεί αυτή η δυνατότητα και ταυτόχρονα να ενδυναμωθεί και ο σύνδεσμος μεταξύ γραπτής δήλωσης και έκθεσης πρωτοβουλίας, με στόχο ενδεχομένω αργότερα να υπάρξει εξέλιξη ή να καταργηθούν τώρα μετατρεπόμενες σε ή μάλλον να, να, να σημειωθεί τώρα ο δεσμός και να μετατρέπονται ορισμένες τουλάχιστον γραπτές δηλώσεις, συγκεκριμένε γραπτές δηλώσεις σε έκθεση πρωτοβουλίας. Και έτσι ίσως κάποιες να είναι και πιο επιτυχείς. Γιατί μπορούμε να πούμε στον κόσμο, ναι, πολύ καλά, όποιες γραπτές δηλώσεις θέλετε, μπορείτε και να τις υποβάλλετε. Αλλά αν δείξετε σοβαρότητα στην υπόθεση αυτή, τότε, αν θέλετε να είσαστε σοβαροί, τότε σκεφτείτε το καλύτερα γιατί θα μπορεί με μία αλφα ε, διαδικασία να μετατραπεί σε έκθεση πρωτοβουλία ή γραπτή δήλωση. Και άρα έτσι δείχνουμε ότι στόχος μας δεν είναι να περιστύλουμε τη δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλία από τους βουλευτές εκείνους που θεωρούν ότι δεν επηρεάζουν ε, την πλειοψηφία ουσιαστικά, αλλά να ε, διαλέξουμε, να επιλέξουμε εκείνες τις πρωτοβουλίες, ε, τις ε, δηλώσεις, οι οποίες είναι ενδιαφέρουσες και σοβαρές και να τις μετατρέψουμε σε εκθέσεις πρωτοβουλίες του Κοινοβουλίου. Αυτά για να συνοψίσω λοιπόν. Το μήνυμα, το δικό μου, και γι' αυτό χρησιμοποιώ και τον όρο καταργείται, καταργηθούν, ήταν να ανακατέψω τα νερά, να προξενήσω συζήτηση, αλλά όπως είπα είμαι υπέρ του εξορθολογισμού, είμαι κατά ιασδήποτε ε, τροπολογίας ισχυρίζεται ότι όλα βαίνουν καλώς με τη γραπτή δήλωση. Γιατί δεν βαίνουν καλώς. Ε, επίσης, ε, όχι στις τροπολογίες εκείνες που λένε ότι θα πρέπει η Επιτροπή να ασχοληθεί με το θέμα κτλ. Ε, ή ότι προσθέτουν μια κάποια αξία. Δεν θέλω να ε, προσβάλλω κανένα, αλλά πρέπει πράγματι να έχει κάποιο νόημα η γραπτή δήλωση. Μπορούμε να προβάλλουμε τους ε, ηλεκτρονικούς τρόπους ε, και να προβάλλουμε την ιδέα της γραπτής δήλωσης γιατί έχει σημασία. Η ιδέα της αδειοδότησης επίσης νομίζω εντάσσεται και αυτή στη λογική του εξορθολογισμού. Και τελευταίο ερώτημα, την ιδέα του Ρομπέρτο με, είτε με τη light εκδοχή είτε με μια πιο συγκεκριμένη διαδικασία πώς θα τη συμπεριλάβουμε στο κείμενο. Αυτό ήταν και το νόημα του αιτήματο για διεύρυνση τη έκθεση μου, έτσι ώστε να μπορεί να φέρει και αλλαγή στι ε, διατάξει. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Thank you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε για την δυνατότητα που έχουμε να συζητήσουμε εις βάθος τις διάφορες εναλλακτικέ για αυτό το ζήτημα. Είναι σημαντικό. Η πρόταση που έκανα αποτελεί αντίδραση σε ένα λεπτό σχόλιο που έγινε από τον Πρόεδρο Κασίνη στην πρώτη μας συνεδρίαση για το θέμα αυτό, ε, ο οποίος ε, έκανε ένα παραλληλισμό αυτού του μέσου με το δικαίωμα πρωτοβουλίας ε, ενός βουλευτή ενός Εθνικού Κοινοβουλίου με τη δυνατότητα να σχετίσει το όνομά του με ένα νομοσχέδιο. Εγώ λοιπόν ε, σκέφτηκα την εξέλιξη του ρόλου του Κοινοβουλίου δυνάμει της Συνδικής της Λισαβόνας και επίσης ε, σκέφτηκα και το ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μία ερμηνεία η οποία ψηφίστηκε από την Επιτροπή αυτή για τον ε, κανόνα 123 και αν η ερμηνεία αυτή ισχύσει θα καταστήσει πιο αυστηρά τα κριτήρια για τη γραπτή δήλωση. Αλλά δεν εφαρμόζεται αυτή η ερμηνεία γιατί θυμάμαι ότι στη σελίδα 74 του εσωτερικού κανονισμού λέγαμε ότι η ερμηνεία λέει το εξή. Το περιεχομένο μια γραπτής δήλωση δεν μπορεί να ε, περβαίνει την επίσημη δήλωση και δεν μπορεί να περιλαμβάνει ένα θέμα λήψη αποφάσεων για το οποίο οι αρμοδιότητε λήψης απόφαση ε, αναγράφονται σε αυτό το εσωτερικό κανονισμό. Έτσι λοιπόν, αυτή η ερμηνεία κατά την άποψή μου θα περιόριζε πάρα πολύ το πεδίο εφαρμογή τη γραπτή δήλωση ε, που αυτή τη στιγμή αντιθέτως εμφανίζεται να γίνεται αποδεκτή. Αποδεκτές για οποιοδήποτε σχεδόν ζήτημα και με οποιαδήποτε μορφή. Συμφωνώ ότι δεν ε, πρέπει να καταργήσουμε την γραπτή δήλωση, αλλά εξορθολογισμό θα μπορούσε να σημαίνει το εξή. Ε, να βάλουμε το πνεύμα τη ερμηνεία αυτή στην πραγματική διαδικασία. Δηλαδή, να περιορίσουμε την ε, δυνατότητα της μη δεσμευτική ε, γραπτής δήλωσης. Γιατί, αν μπορούμε να έχουμε ένα ψήφισμα ή ένα νομοθέτημα, αυτό θα πρέπει να κάνουμε και όχι γραπτή δήλωση αλλά ταυτόχρονα να μην χάσουμε εντελώ το μέσο αυτό, αντιθέτως να το αναβαθμίσουμε, να αναβαθμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο συνδέεται με το άρθρο 42, που είναι το άρθρο για το αποκαλούμενο δικαίωμα πρωτοβουλίας των Ευρωβουλευτών που εφαρμόζουν ε, το άρθρο 125. Έτσι λοιπόν ε, να έχουμε αυτό το άρθρο που να περιορίζει κατά κάποιο τρόπο και να αυξάνει τη δυνατότητα του Προέδρου να μην δέχεται τις περισσότερες από τις γραπτές δηλώσεις, αλλά ταυτόχρονα να μετακινεί και ένα τμήμα αυτών προς ένα πιο σοβαρό μέσο προκειμένου να ενθαρρύνουμε τη χρήση ενός μέσου που τώρα δεν χρησιμοποιούμε ιδιαίτερα. Δηλαδή λέμε ότι έχουμε δικαίωμα πρωτοβουλίας και κανείς δεν χρησιμοποιεί αυτό το δικαίωμα πρωτοβουλίας που έχουμε. Νομίζω ότι καλό θα ήταν, ε, θα άξιζε να πειραματιστούμε. Έτσι λοιπόν δίνοντας την δυνατότητα συλλογής ε, υπογραφών για μία πρόταση για να εκπονηθεί μία έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 225 της συνθήκης θα μπορούσε να υποτελεί αυτό έναν τρόπο αναβάθμισης και ταυτόχρονα θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε και το θέμα της κατάχρησης του μέσου αυτού. Γιατί από ό,τι φαίνεται γίνεται βιομηχανία αυτό με με τα διάφορα λόμπι. Και η κατάσταση που έχουμε σήμερα δεν είναι μια κατάσταση που θεωρώ εγώ ότι είναι αρμόζουσα για ένα κοινοβούλιο που ουσιαστικά θα πρέπει να καταστεί πιο σοβαρό νομοθετικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ λοιπόν τον Ραφαέλ για την ανοιχτή του στάση και ελπίζω ότι και οι υπόλοιποι συνάδελφοι θα το λάβουν αυτά υπόψη. Ευχαριστώ. Κύριος Ντάφ. Ευχαριστώ. Και εμένα μου αρέσει η ιδέα της σύνδεσης, της γραπτής ε, δήλωσης, της διαδικασίας αυτής, προκειμένου να δούμε καλύτερα τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι κάτι που έχουμε παραμελήσει. Μέσω του άρθρου 225. Νομίζω ότι πρέπει να συγχαρούμε τον Ρομπέρτο για το σχέδιο που έχει ετοιμάσει όσον αφορά το άρθρο 42. Θέλω πάντως να βελτιώσουμε την ποιότητα και να μειώσουμε τον αριθμό των γραπτών δηλώσεων. Και αυτό εφαρμόζοντας τα άρθρα του κανονισμού που ήδη έχουμε στη διάθεσή μας. Επίσης, αυξάνοντας και τα κριτήρια προκειμένου να ξεπεραστεί το όριο που έχουμε. Και νομίζω ότι εδώ θα συμφωνήσουμε. Το θέμα είναι να βρούμε το νούμερο, αλλά νομίζω ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ μας ότι πρέπει να γίνει. Τώρα για το τι είναι γραπτή δήλωση. Αν πρέπει να έχει υπεγραφεί πάνω από το 50% των μελών. Τότε έχει και το στοιχείο το ότι είναι δημοφιλής επιπλέον. Δεν πρόκειται μόνο για μια πανηγυρική πράξη. Είναι επίσημη νομοθετική πράξη. Πρέπει να υπάρχει η διάκριση. Μέσω της διαδικασίας αυτής της γραπτής δήλωσης. Μην νομίζουμε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Πρέπει να βρούμε έναν άλλο τρόπο για να το πετύχουμε αυτό. Νομίζω ότι η προσέγγιση του Ρομπέρτο είναι και η σωστή. Συνεπώς, πότε θα ψηφίσουμε, αυτό θέλω να ξέρω. Θα το δούμε αυτό. Εν τω μεταξύ ζήτησε το λόγο ο κύριος Μπρόντς. Ευχαριστώ. Υπάρχουν και άλλες μέθοδοι πρωτοβουλίας για μια πρόταση. Η γραπτή δήλωση έχει το θετικό. Α, αρχίζω να λέω θετικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να σταματήσω τώρα, λέει ο μιλητή. Ε, λοιπόν, έλεγα ότι παραμένει ότι μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι που θα διαφωνήσουν. Πάντως, το θέμα είναι οι προτάσεις που δεν έχουν ε, επιτυχία, που δεν πρόκειται να πετύχουν, πρέπει να δουν το φως της ημέρας παρόλα αυτά κάποια στιγμή. Μήπως τελικά οι απόψεις της μειοψηφίας κάποια στιγμή γίνονται της πλειοψηφίας ή έστω ε, προχωράνε με κάποια συνένεση. Για παράδειγμα, η κατάργηση της θανατικής ποινής στα κράτη-μέλη. Αν ε, τη δεκαετία του 30 ή ακόμα και του 40 και του 50 ρωτούσατε τον κόσμο τι νόμιζε, θα βλέπατε ότι πολύ λίγοι θέλανε την κατάργηση. Και θα λέγαμε ότι ήταν και πολύ ε, περίεργη η άποψή τους. Όμως σιγά σιγά έγινε ε, συνένεση. Νομοθετικά τουλάχιστον υπάρχει αυτή η συνένεση. Τώρα, ε, χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο είχαν τον είχαν κανόνες που ήταν τις μειοψηφία κάποια στιγμή, με τα επιχειρήματα αλλάζει η κατάσταση. Το ίδιο θέλω να πω και για την γραπτή δήλωση. Μπορεί να ξεκινάει σαν μία μειοψηφική άποψη, να ακούγεται τρελή, υπερβολική, αλλά σιγά σιγά ακούγεται το επιχείρημα και ο κόσμος έτσι έχει την ευκαιρία να το δεχτεί ή να μην το δεχτεί. Αυτό θέλω να πω για την γραπτή δήλωση για τις γραπτές δηλώσεις με στήριξη της πλειοψηφίας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει νομοθετικό κύρος και άρα δεν μπορεί να είναι δεσμευτική, κατά τη γνώμη μου. Αυτό θέλω να πω. Πριν να ξαναδώσουμε το λόγο στον συνάδελφο Ταρκόφσκι να απαντήσει, ευχαριστώ τον κύριο Γκολτιέρη που αναφέρθηκε στις παρατηρήσεις του παρελθόντος. Ε, όμως, αυτά που είπαμε στο παρελθόν ε, εκφράζουν ένα συνέστημα, αλλά ε, αυτό το να προχωρά κάποιος στους διαδρόμους και να υπάρχουν διάφορα άτομα που προσφέρουν φυλάδια δεν νομίζω ότι είναι μια εικόνα που ανταποκρίνεται στη σοβαρότητα που πρέπει να έχει ο οίκος αυτός, όμως ε, πολλές φορές ε, γράφονται κάποιες τέτοιες ε, δηλώσεις για να ικανοποιήσουμε την κοπελίτσα που δίνει το φυλάδιο. Έτσι λοιπόν δεν ξέρω, ίσως θα έπρεπε να αποφευχθεί κάτι τέτοιο και νομίζω ότι πρέπει να αυξηθεί η σοβαρότητα. Λοιπόν, ο εισηγητή έχει το λόγο. Δεν έχω πολύ χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω πολλά να πω μάλλον. Ε, θα προσπαθήσουμε να βρούμε συμβαστικές λύσεις. Είπαμε ότι πρέπει απλώ να μελετήσουμε πιο προσεκτικά την πρόταση του Ρομπέρτο για να τη διευκρινίσουμε στα άλλα ζητήματα μπορούμε νομίζω εύκολα να βρούμε συμβαστικέ λύσεις. Στην πρώτη, του Ρομπέρτο θα πρέπει να δουλέψουμε λίγο πιο προσεκτικά για να βρούμε μία απόλυτα καλή και στεγανή, ε, άψογη δηλαδή λύση. Για το χρονοδιάγραμμα ίσως μπορεί να μας βοηθήσει η γραμματεία τι πρόγραμμα έχει. Μου προτείνει η γραμματεία να προτείνουμε τη 30 Μαΐου. 30 Μαΐου για το θέμα αυτό. Η ψηφορία συμφωνείτε. Αυτό σημαίνει ότι οι τροπολογίες μπορούν να κατευθούν μέχρι τις 29. Εκτός μικροφώνου τα σχόλια του κ. Κολτιέρη. Λοιπόν, αν μπορούσατε να το κάνετε τον Ιούνιο θα ήταν καλύτερο να έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο. Αυτή ήταν η πρόταση της γραμματείας. 15 Ιουνίου, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, απλώς να σας υπενθυμίσω ότι η επόμενη συνεδρίαση θα λάβει χώρα στις 29 Μαΐου από τις 3 ω τις 6.30 εδώ στις Βρυξέλλες, Τρίτη και κατόπιν Τετάρτη, 30 Μαΐου από τι 9 το πρωί ως τις 12.30 πάλι στις Βρυξέλλες. Ολοκληρώνεται εδώ η συνεδρίασή μας. Σας ευχαριστώ Σε όσους είχατε την υπομονή να μείνετε μέχρι το τέλος.